Καλησπέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στην συνεδρίαση της Επιτροπής Βιομηχανίας Έρευνας και Ενέργειας. Αν δεν υπάρχουν ε, παρατηρήσεις μπορούμε να εγκρίνουμε τη μερίστη διάταξη χωρίς καμία τροποποίηση. Δεν νομίζω ότι θέλει να πάρει κανείς το λόγο. Παρατηρήσεις παρακαλώ. Όχι. Περνάμε στο σημείο 2 της ημερήσιας διάταξης, ανακοινώσει του Προέδρου. Κάτι πολύ σημαντικό. Η αυριανή συνεδρίαση τη Επιτροπή μα αύριο το απόγευμα θα ξεκινήσει στι 4 παρατέταρτο, 15 και 45. 4 παρατέταρτο. Όχι στι 3 λοιπόν ω ήθιστε, αλλά στι 4 παρατέταρτο και θα λάβει χώρα σε διαφορετική αίθουσα συνεδριάσεων, συγκεκριμένα στην Paul Ενρίς Πακ 5Β001. στον πέμπτο όροφο δηλαδή αυτού του κτηρίου. Εκεί θα διεξαχθεί η αυριανή απογευματινή μα συνεδρίαση. Περνάμε στο σημείο 3 τη ημερήσια διάταξη, μελέτη με θέμα τη επενδύση στην Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Βιομηχανία, παρουσίαση από του Λουκ Νούφελ και την Τζέσικα Γιερουντ. Να καλωσορίσω καταρχά του δύο εμπειρογνώμονε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σα ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σα εδώ. Η μελέτη αυτή προτιμάστηκε από την εταιρεία Trinomics, που είναι ένα γραφείο παροχής συμβουλών στο τομέα της οικονομικής πολιτικής μέτρα το Ρόντερταμ, που διεξάγει έρευνα και παρέχει συμβουλές χάραξης πολιτικής στο τομέα της ενέργειας, του περιβάλλοντος και των κλιματικών αλλαγών, τομείς που είναι πάρα πολύ σημαντική για την Επιτροπή μας. Οι δύο λοιπόν προσκεκλημένοι μας, ο κύριος Λουκ Βαν Νούφελ η κυρία Τζέσικα Γίργουτ βρίσκονται εδώ πέρα. Ο κύριο Βαν Κνούφελ εργάζεται το 2015 στην ε, Trinomics, το ίδιο και η Τζέσικα Γίργουτ, η οποία είναι σύμβουλο στον τομέα τη ενέργειας στην ε, Trinomics. Η κυρία Γίργουτ ασχολείται με, με τα θέματα της βιώσιμης ενέργειας, της, ε, βιώσιμης, της χρηματοδότησης μάλλον της βιώσιμης ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης και της διακυβέρνησης στον τομέα της ε, ε, ενέργειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο κύριος Γκλουκ Βανούφελ με τη σειρά του ασχολείται ιδιαίτερα με τον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου στο Βέλγιο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο Έχει παράσχει συμβουλές σε οργανισμούς όπως ε, η Παγκόσμια Τράπεζα, ο Φλαμαδικός Οργανισμός Ηλεκτρικής Ενέργειας, καθώς επίσης και στην ε, Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση του Βελγίου. Σας καλωσορίσουμε λοιπόν και τους δύο. Και πρέπει να σας πω ότι ε, οι δύο καλεσμένοι μας έχουν αναλύσει τις εκτιμόμενες επενδυτικές ανάγκες, καθώς επίσης και τα κίνητρα αλλά και τα εμπόδια στον τομέα των επενδύσεων όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια με βάση τα διάφορα τεχνολογικά σενάρια τα οποία απαιτούνται προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι, οι ενεργειακοί και οι στόχοι αντιμετώπισης κλιματικής αλλαγής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρετε αυτή τη στιγμή ότι ε, ασχολούμαστε ιδιαίτερα με το ζήτημα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και ενός νέου μοντέλου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και πώς θα μπορούσαν να σχεδιαστούν οι σχετικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας. Εσείς κάνετε μια αξιολόγηση διαφόρων πιθανών επιλογών πολιτικής προκειμένου να προωθηθούν οι απαραίτητες επενδύσεις στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και πραγματικά χρειαζόμαστε τέτοιες αναλύσεις και τέτοιες συστάσεις στον τομέα αυτό. Είναι πραγματικά σημαντικό για μας να δούμε Πώ έχουν τα πράγματα, πώ τα βλέπετε εσεί που είστε επαγγελματίε και πυρογνώμονε, ποιε συμβουλέ μπορείτε να μα δώσετε προκειμένου να διαμορφωθεί καλύτερα ο τομέας αυτός. Πώς μπορεί δηλαδή να ρυθμιστεί ο κλάδος αυτός με ένα καλύτερο τρόπο. Οι νουθυσίες αυτές είναι πολύ σημαντικές προκειμένου να καταφέρουμε να προωθήσουμε και συγκεκριμένα νομοθετήματα, όπως για παράδειγμα το ζήτημα της διακυβέρνησης, του σχεδιασμού της αγοράς, τι θα γίνει με τους ε, Acer, με, τους, ε, με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Όλα αυτά μπορούν να εμπλωτιστούν περισσότερο με τις δικές σας συμβουλές, με τη δική σας την ανάλυση. Να ζητήσω καταρχάς από τον κύριο Λουκ Βανούφελ να πάρει το λόγο. Ή η κυρία Γέργουτ, μάλλον. Η κυρία Τζέσικα Γέργουτ, λοιπόν, έχει το λόγο. Θα... Νομίζω ότι ακολουθούσα αλφαβητική σειρά, αλλά δεν ακολουθούμε αλφαβητική σειρά. Η κυρία Γέργουτ, λοιπόν, έχει το λόγο. Σας Ευχαριστώ πολύ για, την, ε, για τα ζωικά σε αυτά λόγια. Όντω θέλουμε αυτή τη στιγμή να δούμε μέσω τη μελέτη αυτή πώ μπορούμε να διευκολύνουμε περισσότερο τι επενδύσει στον τομέα τη ηλεκτρική ενέργεια, προκειμένου να επιτευχθεί η μετάβαση σε έναν ενεργειακό εφοδιασμό χαμηλών εκπομπών άνθρακα μέχρι το 2050. Προκειμένου να γίνει αυτό, έχουμε εξετάσει διάφορε πτυχέ του ζητήματο ασχοληθήκαμε καταρχάς με τους στόχους ενεργειακής πολιτικής και της πολιτικής για την αλλαγή του κλίματος. Είδαμε επιδείσεις ποιες επενδύσεις απαιτούνται προκειμένου να επιτύχουμε τους στόχους αυτούς. Κάναμε μια ανάλυση των ευρωπαϊκών μέσων προκειμένου να δούμε ποιες είναι οι επενδύσεις και πώς μπορούν να ρυθμιστούν και πώς μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Είδαμε επίσης ποιε είναι οι διάφορες επενδυτικές τάσει, οι φραγμοί, τα εμπόδια αλλά και οι κινητήριες δυνάμεις για τι επενδύσει αυτέ. και καταλήγουμε στο τέλος σε πιθανές επιλογές χάραξης πολιτικής και σε κάποιες συστάσεις. Προκειμένου να γίνουν όλα αυτά, χρησιμοποίησαμε μια εκτεταμένη βιβλιογραφία και κάναμε και τρεις περιπτωσιολογικές μελέτες για τρεις συγκεκριμένε περιοχές και ήρθαμε σε επαφή και με διάφορους ενδιαφερομένους. Ξεκινώντας λοιπόν θελήσαμε να εντοπίσουμε τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής και της πολιτικής για την πενόπιση των κλιματικών αλλαγών. Τα τελευταία χρόνια προσπαθούμε να λύσουμε ένα τρίλημα, όπως βλέπετε εδώ πέρα, μια επιλογή ανάμεσα σε τρεις εναλλακτικέ. Να καταφέρουμε να κάνουμε καταρχάς πιο ασφαλή, πιο βιώσιμη και πιο ανταγωνιστική την, τον εφοδιασμό των ενεργειακών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό το λόγο θέσαμε διάφορους στόχους. Στόχους 2020 και 2030 όσον αφορά το κλιματολογικό πλαίσιο. Έχουμε συγκεκριμένους στόχους εδώ πέρα για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, για την ενεργειακή απόδοση και την ενεργειακή διασύνδεση, καθώς επίσης και την ευφυή μέτρηση. Με τις υφιστάμενες αυτές τάσεις βλέπουμε ότι τα περισσότερα κράτη-μέλη ευθυγραμμίζονται για την επίτευξη των στόχων του 2020, χρειάζονται όμως περαιτέρω επενδύσεις και περαιτέρω διαμόρφωση πολιτικής για να πετύχουμε τους στόχους του 2030 και του 2050. Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι με χρονικό ρίστο το 2050, θα πρέπει να έχουμε μια σημαντική μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, και γι' αυτό το λόγο χρειαζόμαστε και πάρα πολύ σημαντικέ επενδύσει στον τομέα παραγωγή ηλεκτρική ενέργεια. Θα έλεγα ότι οι πιο σημαντικέ επενδύσει είναι στην παραγωγή ηλεκτρική ενέργεια, 54 με 80 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίω μέχρι το 2050, εκ των οποίων περίπου 75 με 80% θα έχουν να κάνουν με τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Και έπειτα για τα ηλεκτρικά δίκτυα 40 με 62 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως θα πετηθούν μέχρι το 2050 εκ των οποίων περίπου ένα 80% απαιτούνται για τα δίκτυα δια... διανομής. Και κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να καλύψουμε και την συμπαραγωγή σε μικρή κλίμακα, αλλά και την παραγωγή ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιεί ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Επίση, είναι σημαντικό να δούμε τι γίνεται στον τομέα τη διασύνδεση, καθώ επίση και στον τομέα τη αποκατάσταση, επισκευή και ανανέωση των δικτύων. Και έχουμε και το ζήτημα τη αποθήκευση, καθώ επίση και τι επενδύσει πρέπει να γίνουν για να αποκριθούμε στη ζήτηση. Οι επενδύσει εδώ πέρα είναι χαμηλέ, αλλά πιστεύω θα αυξηθούν στο μέλλον. Απαιτούνται λοιπόν επενδύσεις προκειμένου να πετύχουμε τους στόχους του 2050 για τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα και γι' αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιεί διάφορα εργαλεία. Από ρυθμιστικής πλευρά θα έλεγα ότι τα πιο σημαντικά είναι τα ευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα της ενέργειας, ένας κανονισμός συγκεκριμένα που περιέχει και ένα πλαίσιο για τα σχέδια κοινού ενδιαφέροντος. Έχουμε επίσης την οδηγία για τι ανώσιμες πηγές ενέργειας και το σύστημα Εμπορίε εκπομπών. Υπάρχουν όμω και διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω η διευκόλυνση συνδέοντα στην Ευρώπη, που υποστηρίζει σχέδια κοινού ενδιαφέροντο. Έχουμε τον ΕΡ 300, τον Ορίζοντα 2020, όπου επικεντρώνονται περισσότερο στην κοινοτομία και την έρευνα. Και έχουμε και κάποια γενικότερα, αν θέλετε, ταμεία, όπω το ΕΦΣΙ και το ΕΣΥΦ, τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Τα χρηματοδοτικά αυτά μέσα παρέχουν περίπου 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως σε επιδοτήσεις και 12,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε χρηματοδοτικά μέσα για όλα τα σχέδια του ενεργειακά, που αντιστοιχούν όμως μόνο στο 10 με 15% των ετήσιων επενδυτικών αναγκών που έχουμε εντοπίσει μόνο και μόνο για τον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι χρειάζονται και περαιτέρω χρηματοδοτήσεις στον τομέα αυτών. για να παρουσιάσουμε τώρα κάποιες από τις επενδυτικές στάσεις που έχουμε εντοπίσει όσον αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Θα ξεκινήσω με την παραγωγή ενέργειας με βάση τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ο συνάδελφός μου έπειτα θα συνεχίσει με τις υπόλοιπες συναδειόμενες στάσεις. Όσον αφορά λοιπόν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έχουμε εντοπίσει ότι το κόστος εδώ πέρα μειώνει όλο και περισσότερο και ότι κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να προωθήσουμε περισσότερο τις επενδύσεις αυτές σε σχέση με τη συμβατική παραγωγή. 50 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2015 ήταν οι επενδύσεις στον τομέα αυτών. Και έχουμε εξαπλάσια λοιπόν αύξηση των επενδύσεων σε σχέση με το 2004. Το 2004 η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν στην πρώτη γραμμή όσον αφορά τις νόσιμε πηγές ενέργειας, Τώρα η Κίνα βρίσκεται στην πρώτη θέση. Ωστόσο, οι επενδύσει αυτέ δεν είναι ισότιμα κατανεμημένε σε όλα τα κράτη-μέλη. Υπάρχουν μεγάλε αποκλήσει από το ένα κράτο μέλο στο άλλο και βασίζονται ακόμα πολύ σε επιδοτήσει. Μολονότι μειώνονται οι επιδοτήσει αυτέ ανά μεγαβατόρα, αρχίζουν και βασίζονται όλο περισσότερο σε πραγματικές συνθήκε αγορά. Όσον αφορά τώρα την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στη συμβατική, εδώ είδαμε ότι όλο και δυσδύουν περισσότερο ενενώσιμες πηγές ενέργειας, πράγμα το οποίο έχει πειράσει την κερδοφορία των συμβατικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και βλέπουμε ότι όλο και περισσότερο οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας που χρησιμοποιούν πυρηνική ενέργεια, ορυκτά καύσιμα, παροπλίζονται ουσιαστικά και τίθενται οριστικά εκτός λειτουργίας. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ακόμα ένα επιχειρηματικό μοντέλο συγκεκριμένο με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλά κράτη-μέλη τα οποία χρησιμοποιούν μηχανισμούς χρηματοδότησης των ικανοτήτων ηλεκτροπαραγωγής προκειμένου να αντισταθμίσουν την ε, όλο και μεγαλύτερη μείωση της χρησιμοποίησης των συμβατικών μορφών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι ε, οι ανανόσιμες πηγές ενέργειας χρηματοδοτούνται όλο και περισσότερο, προωθούνται όλο και περισσότερο από την πολιτική την οποία ακολουθούμε, αλλά χρειάζονται παρόλα αυτά πάρα πολλέ επενδύσει προκειμένου να καταφέρουμε να αποκαταστήσουμε κάποιε παροχημένε μονάδε παραγωγή ηλεκτρική ενέργεια. Βλέπουμε ότι αυξάνονται όλο και περισσότερα τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία επηρεάζονται και αυτά από τη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αυτό το βλέπουμε στο μείγμα ηλεκτρικής παραγωγής όπου είναι 38% αντιστοιχεί στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Βλέπετε εδώ πέρα ποια είναι η κατανομή μεταξύ ολικής ενέργειας, ηλιακής ενέργειας και άλλων μορφών ενέργειας όπου το μείγμα αυτό είναι ιδιαίτερα υψηλό σε χώρες όπως η Γερμανία. Θα λέγαμε λοιπόν ότι μέχρι στιγμή δεν έχουμε εντοπίσει προβλήματα όσον αφορά τη δυνατότητα λειτουργία του συστήματο και των δικτύων διανομή ηλεκτρική ενέργεια με τη χρησιμοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργεια. Αν όμω αρχίσει και αυξάνεται το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια, θα πρέπει να προσαρμόσουμε την ισορροπία της χρησιμοποίησης διαφορετικών πηγών ενέργειας. Αυτή τη στιγμή χρειάζεται λοιπόν μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά την ε, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θα πρέπει παράλληλα να προβλεφθούν και απαραίτητα μέτρα τόσο για την αποθήκευση ενέργειας όσο και για την ε, ανταπόκριση στην αυξανόμενη ζήτηση. Αυτό είχε γίνει στο παρελθόν με συγκεκριμένες συμβάσεις από τη βιομηχανία και τώρα βλέπουμε ότι καλύπτει όλο και περισσότερο την παροχή ενέργειας προς τους πολίτες, προς κατοικίες. Όσον αφορά τώρα την αποθήκευση, εδώ πέρα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν συγκεκριμένες τεχνολογίες οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές και πολλές φορές αντιστοιχούν ακόμα και στο 95% της αποθήκευσης στην Ευρώπη. Όλο και νέες τεχνολογίες όμως αναπτύσσονται αυτή τη στιγμή όπως η τεχνολογία Patris, η οποία χρησιμοποιείται στη Γερμανία σε ένα ποσοστό 40%. Βλέπουμε ότι ε, υπάρχουν όλο και περισσότερες εγκαταστάσεις στη Γερμανία που χρησιμοποιούν ε, στήλες εισόρευσης προκειμένου να αποθηκεύεται όλο και περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια. Αυτό σε συνδυασμό με τη γενικότερη τάση ψηφιοποίησης του τομέα αυτού μπορούμε να πούμε ότι αλλάζει εντελώ το τοπίο και το περιβάλλον όσον αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και όσον αφορά τις υπηρεσίες αυτές που παρέχουν ε, οι φορείς εκμετάλλευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό λοιπόν επίσης είναι πολύ σημαντικό στοιχείο στην ε, εξέλιξη του τομέα ενέργειας. Η διείσδυση των ανανεώσιμων και οι άλλες επενδύσεις οδηγούν σε αύξηση του λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό πρέπει οπωσδήποτε να ληφθεί υπόψη, ε, δηλαδή κατά πόσον είναι οι οικονομικές οι λύσεις το κόστος του συστήματος το 2030 θα είναι περίπου αυξημένο κατά 30% σε σχέση με το 2010. Παρά τις χαμηλότερες τιμές χονδρικής, ή συνολικές, τα συνολικά κόστη για την ενέργεια αυξάνονται. Όλοι γνωρίζομαι δύο άλλες τάσεις στον τομέα ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή εξηλεκτρισμός μεταφορών και θέρμανσης. μεταφορές, εκεί υπάρχει μια διείσδυση 80% αναμενόμενη διείσδυση το 2050. Ο αντίκτυπος θα είναι πολύ μεγάλος. Τώρα είναι περίπου το 10% της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και 150 ΜΒ δυνατότητα παραγωγής, ικανότητα παραγωγής ενέργειας. Ο εξηλεκτρισμός στον τομέα της θέρμανσης είναι αρκετά καινούριο, με αντλίες θερμότητας για παράδειγμα, με εσωτερικά πάνελ, με θερμικά πάνελ. Ε, έχουμε δει στον τύπο ότι στην Ολλανδία για παράδειγμα η κυβέρνηση πήρε μια στρατηγική απόφαση να σταματήσει την χρήση αερίου σταδιακά για λόγους θέρμανσης και καταρχήν δεν θα συνεχιστούν, δηλαδή για τη θέρμανση δεν θα, γίνουν πια, δεν θα γίνονται πια επενδύσεις στο αέριο. Υπάρχει πολύ μεγάλη οικονομική υποστήριξη για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και χρήση ηλεκτρικής ενέργειας. Ε, είναι πολύ μεγάλη η αύξηση εδώ από το 2008 μέχρι το 2012. Η αύξηση δεν είναι μόνο σημαντική για τις ανανεώσιμες πηγές 90% αλλά και για τα ορυκτά καύσιμα 39%. Είναι μάλλον περίεργο ότι τα ορυκτά καύσιμα και άνθρακας δηλαδή και φυσικό αέριο ακόμα επιδοτούνται σε σημαντικό επίπεδο. Και αυτή είναι μία από τις συστάσεις μας δηλαδή σταδιακή αντικατάσταση αυτών των πηγών ε, ενέργειας. Για να περάσουμε σε αυτή τη φάση μετάβασης ε, ενέργειας χωρίς ε, πολυάνθρακα. Ξέρω τα καινούρια χρηματοδοτικά μέσα, δηλαδή τοπικές συμπράξεις, ε, που συνεργάζονται ε, τώρα δηλαδή χρηματοδοτούνται τα έργα και υπάρχουν και ιδιωτικά ίδια κεφάλαια και τοπική συμμετοχή. Τώρα, ποιες, ε, ποιοι είναι οι προωθητικοί παράγοντες και τα εμπόδια, τα βασικά. ιστορικά η αύξηση της ενέργειας ήταν ένα, μια, ένας προωθητικός παράγοντας. Τώρα όμως αυτό έχει περιοριστεί. Η περισσότερη ανάπτυξη στον τομέα της ενέργειας καλύπτεται από επενδύσεις στα ανανεώσιμες πηγές. Τα επίπεδα απολαβών, ε, η Τζέσικα το είπε, είναι αρκετά χαμηλά. Αυτό δεν είναι εμπόδιο λοιπόν. μπορούμε να εστιάσουμε στα πιο σημαντικά υπέρ και κατά για να σεβαστούμε και το χρόνο και εδώ πρέπει να πούμε ότι ο βασικότερος προθετικός παράγων στην αγορά σήμερα είναι η υποστήριξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ε, ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια είναι ε, η διαδικασία αδειοδότησης και η έγκριση των υποδομών γενικότερα. Αυτά είναι κρίσιμα θέματα και στη σημερινή κατάσταση. Και η δημόσια αποδοχή των υποδομών. Ε, έχουμε εξετάσει θεωρητικά 12 πολιτικές επιλογές. Η πρώτη ομάδα επικεντρώνεται στη λειτουργία των αγορών η δεύτερη ομάδα, στη δεύτερη ομάδα έχουμε εντοπίσει πολιτικές επιλογές που θα καταστούν αναγκαίες αν δεν λειτουργεί σωστά η αγορά και η τρίτη ομάδα πολιτικών επιλογών αφορά το γενικότερο ρυθμιστικό πλαίσιο. Και το συμπέρασμά μας είναι ότι οι πολιτικές επιλογές που θέλουν να βελτιώσουν τη λειτουργία της αγοράς είναι οι αποδοτικότερες και οι καταλληλότερες. Γιατί αντιδρούν σωστά στα διάφορα κριτήρια και αποκρίνονται στα κριτήρια που έχουμε ε, θέσει για να αξιολογήσουν τις διάφορες πολιτικές επιλογές. Ταξινομήσαμε τις διάφορες πολιτικές επιλογές λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπό τους και παρουσιάσαμε εδώ τις θετικότερες έξι επιλογές. Αυτά τα συμπεράσματα βέβαια ε, αναφέρονται και στις συστάσεις, μεταφέρονται και εκεί. Προτείνω λοιπόν να περάσουμε στις συστάσεις που είναι το σημαντικότερο κομμάτι της μελέτης μας βέβαια. Η πρώτη σύσταση εστιάζει στην ανάγκη επενδυτικής ασφάλειας βεβαιότητας. Αυτό είναι ένα μήνυμα που επαναλαμβάνεται σε διάφορες μελέτες αλλά και μηνύματα που παίρνουμε από τη βιομηχανία. Η ε, ασφάλεια των επενδυτών είναι κλειδί για όλες τις επενδύσεις, όχι στα δίκτυα, όχι μόνο στην παραγωγή ενέργεια, αλλά ε, και σε συμβατικές ε, μεθόδους κλπ. Είδαμε στη ε, περίπτωση μελέτης για την Ισπανία η πολιτική για τα αναλώσιμα άλλαξε το 2013 με αναδρομική ισχύ και αυτό οδήγησε σε πάγωμα όλων των επενδύσεων. Οπότε αυτό είναι κέριο ζήτημα. Δεύτερον, οι ανανεώσιμες πηγές θα πρέπει να στηρίζονται με τρόπο σταθερό και προβλέψιμο, αυτό έχει σχέση με την πρώτη σύσταση βέβαια, αλλά και ολόκληρη υποστήριξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να είναι πιο συντονισμένη μεταξύ των κρατών μελών σε περιφερειακό επίπεδο και να στηρίζεται περισσότερο στην αγορά. Οι πρόσφατες εξελίξεις νομίζω ότι πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση στην ε, διαδικασία διαγωνισμών που θεσμοθετήθηκε, αυτό είναι καλό, και υπάρχουν και νέες προτάσεις στο, στο χειμερινό πακέτο ε, που είναι θετικές. Είναι καλά βήματα για την έρευνα και την ανάπτυξη σημειώνουμε ότι οι προσπάθειες έρευνας και ανάπτυξης είναι θετικές και σωστές. Ποσοτικά, δηλαδή η Ευρώπη επενδύει όσο πρέπει για την ενέργεια και τις ανανεώσιμες πηγές, αλλά υπάρχει ακόμα περιθώριο βελτιώσεων, δηλαδή καλύτερος συντονισμός και στις νέες τεχνολογίες, ε, νέα αντιλήψεις και μοντέλα αγοράς κλπ. Η ασφάλεια του εφοδιασμού είναι ένα άλλο σημαντικό θέμα της προσφοράς και εδώ επαναλαμβάνουμε τη σύσταση ότι οι πρωτοβουλίες των κρατών μελών θα πρέπει να συντονίζονται περισσότερο σε περιφερειακό επίπεδο και οι δυνατόν και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, σε ό,τι αφορά την αποθήκευση υπάρχει ε, ανάγκη ε, εναρμονισμένου ρυθμιστικού πλαισίου σε επίπεδο ένωσης και αυτή είναι μια ιδέα που περιλαμβάνεται στο χειμερινό πακέτο. Και η τελευταία σύσταση στην πρώτη ομάδα έχει να κάνει με την ικανότητα διασύνδεσης. Χαιρετίζουμε το στόχο που έθεσε ε, ο Ευρωπαίος Νομοθέτης το 10% αλλά πιστεύουμε ότι ε, ε, ένας στόχος διαφοροποιημένος θα ήταν καταλληλότερος. Και εκείνοι που χαράζουν την πολιτική θα πρέπει να εστιάζουν στη διαθεσιμότητα της ικανότητας παραγωγής. Όχι μόνο την ε, φυσική διαθεσιμότητα παραγωγής ενέργειας, αλλά αυτή η φυσική ικανότητα θα πρέπει να διατίθεται στην αγορά. Και αυτό είναι ένα κρίσιμο ζήτημα σήμερα. Μια άλλη σύσταση εστιάζει στην ανάγκη κατάλληλου ρυθμιστικού πλαισίου για τις επενδύσεις και βέβαια αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ε, παρέχονται κίνητρα για αυτούς που χειρίζονται, διαχειρίζονται και λειτουργούν τα δίκτυα, αλλά και στο σκέλος της προσφοράς. Η πρόσβαση ε, σε συγχρηματοδότηση, σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, σε εταίρους είναι σημαντικό θέμα. Πολλά έχουν επιληθεί, αλλά υπάρχουν ορισμένε λεπτομέρειες που θέλουμε να προσθέσουμε, όπως η πρόσβαση στα ε, χρηματοδοτικά μέσα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να διευκολύνεται χωρίς επικαλύψεις και μικρότερα έργα και μικρότεροι διαχειριστές θα πρέπει να είναι επιλέξιμοι για χρηματοδότηση. Και αυτό να γίνεται ε, συνενώνοντας ε, πρωτοβουλίες. Οι τιμές είναι πολύ σημαντικές, χρειάζεται σωστή τιμολόγηση για την ηλεκτρική ενέργεια, για τον άνθρακα και τα δίκτυα. Ε, νομοθετικά ρυθμιζόμενες ε, ε τιμές ε, δεν είναι πλέον προωθητικός παράγων και θα πρέπει να καταργηθούν. Αυτό έχει γίνει αναγκαιότητα και προτεραιότητα για να δοθούν κίνητρα για τις επενδύσεις οι τιμές σήμερα είναι χαμηλές, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη αυτό. Πρέπει δηλαδή να ληφθούν μέτρα αύξησης των τιμών. Για την ε, ενεργειακή απόδοση, εδώ εστιάζουμε στην ανάγκη κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου, ρυθμιστικού πλαισίου και εδώ χρειάζονται πρωτοβουλίες σε ενωσιακό επίπεδο, ούτω ώστε να οριστούν οι αρμοδιότητες, ε, κάποιοι κανόνες εις ό,τι αφορά την ιδιοκτησία δεδομένων, την επικοινωνία κλπ. Τέλος, εις ό,τι αφορά την αδειοδότηση, οι διαδικασίες θα πρέπει να απλουστευθούν, να γίνουν συντομότερες και η δημόσια αποδοχή, η αποδοχή από το κοινό είναι ένα θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει περισσότερο. Υπάρχουν κάποιες ιδέες, κάποιες βέλτιστες πρακτικές, οι επενδυτές και οι αρχές θα πρέπει να ενημερώνουν το κοινό σε εκδηλώσεις και θα πρέπει να προσφέρουν πρόσβαση ε, στα έργα τα χρηματοδοτούμενα και συγχρηματοδοτούμενα μέσα από, συνεργαζόμενες, από, από συνεργατικές συμπράξεις. Αυτή είναι πραγματικότητα σήμερα σε κάποια κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορούν να θεωρηθούν αυτά βέλτιστες πρακτικές για όλα τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και είμαστε στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση αυτή και η ε, έκθεσή σας είναι πολύ σημαντική για μας. Ο συνάδελφος Λεβαντόφσκι. Ευχαριστώ, συμφωνώ ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η έκθεση και φιλόδοξες και οι συστάσεις. Δύο σύντομες ερωτήσεις. Στη μελέτη σας ε, Κάνετε μια εκτίμηση σε αιτήσια βάση αυτού που χρειάζεται και λέτε πάνω από 140 δις ευρώ για παραγωγή ενέργειας και διανομή. Μεταφορά. Πολύ περισσότερο από την ικανότητα που έχουν όλα τα μέσα της Ένωσης. Πριν από δύο εβδομάδες ψηφίσαμε την ε, αναθεώρηση του συστήματος εμπορίας εκπομπών θεωρήσαμε ότι ε, θα έπρεπε να αυξηθεί η τιμή των δικαιωμάτων. Εσείς πώς βλέπετε την, τον αντίκτυπο α, της αύξησης ε, των δικαιωμάτων εκπομπών ε, διοξιδίου του άνθρακα σε σχέση με τις επενδύσεις που χρειάζονται για να επιτευχθούν οι φιλόδοξοι στόχοι. Δεύτερον, μια ερώτηση για τις επιχειρήσεις και το προφίλ κινδύνου και του τι πρέπει να χρηματοδοτεί το ΕΦΣΙ, το έτσι και ο Ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός. Ε, δηλαδή στον ενεργειακό τομέα αναχώρα τι θα επενδύσεις θα γίνουν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριος Μάιερ. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ για την παρουσίαση. Μια ερώτηση έχω, ειδικότερα για τις επενδύσεις στα δίκτυα. Στην παρουσίασή σας δεν μας είπατε για την αποκεντρωμένη παραγωγή ενέργειας Βέβαια θεμητό, γιατί δεν ξέρουμε ποιο μοντέλο θα υπερισχύσει. Αλλά στο μέλλον θεωρούμε ότι η αποκεντρωμένη παραγωγή θα παίξει ρόλο σημαντικό. Αυτή η παραγωγή όμως, όπως λέμε, δεν χρειάζεται ε, ευρύ δίκτυο, εκταταμένο δίκτυο. Αν ισχύει αυτό, πώς θα γίνουν οι επενδύσεις ε, στο δίκτυο. Δηλαδή, μπορεί να γίνει συνδυασμός ε, δικτύων και συστημάτων αποθήκευσης ή υπάρχει κίνδυνος αν αυξηθούν οι επενδύσεις στα δίκτυα να είναι επενδύσεις που θα αυξήσουν μόνο το κόστος της ε, ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς να έχουν ε, απόδοση. Ευχαριστώ, συνάδελφες Κρούλετ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είδα στην παρουσίασή σας ότι αναφέρατε το ΚΑΠΕΚ σε μια διαφάνεια. Δηλαδή κόστος κεφαλαιοχικής επένδυσης στα κράτη-μέλη. Υπάρχουν δεδομένα γι' αυτό, γιατί ξέρω ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ αναπτυγμένων και λιγότερο αναπτυγμένων κρατών μελών. Ε, δηλαδή, πώς θα γίνουν οι επενδύσεις στην ίδια τεχνολογία. Υπάρχει εδώ μια ανισότητα σε μη αναπτυγμένα κράτη-μέλη. Υπάρχουν μεγαλύτεροι κίνδυνοι. Και το, ε, οι επενδυτικές ανάγκες ως προς το κόστος είναι υψηλότερες από τις αναπτυγμένες χώρες. Δεύτερον, μια ερώτηση για την ευελιξία. Είδα και το κείμενό σας στη μελέτη. Ε, ε, είπατε λίγα πράγματα για την αποθήκευση και ε, υπάρχει σύσταση σε σχέση με την ανάπτυξη της τεχνολογίας αποθήκευσης στις ΙΠΑ, στην Κίνα. Ήδη ε, έχουν τεράστια αποθηκευτική ικανότητα. Ε, εμείς ε, εδώ έχουμε ένα πρόβλημα. Δηλαδή, ε, ακόμα ε, μιλούμε θεωρητικά για το θέμα αυτό της αποθήκευσης ενέργειας. Τέλος, τεχνολογίες ε, πληροφορίας και επικοινωνίας. Τεχνο, τεχνολογίες πληροφορίας, που θα επιτρέψουν μεγαλύτερη συμμετοχή από το κοινό πώς επηρεάζει η τεχνολογία της πληροφορίας ε, το επόμενο διάστημα μέχρι το 2030. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. να σας θέσω και εγώ μια-δύο ερωτήσεις. αν κατάλαβα καλά τα όσα είπατε, η πρόσβαση στη χρηματοδότηση δεν είναι πρόβλημα. Πολύ αισιόδοξο σας βρίσκω αυτή τη δήλωση. Πολύ μου άρεσε. Αλλά τι γίνεται με τον μηχανισμό ανάπτυξης δυνατοτήτων. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε αρκετές επενδύσεις και κανείς δεν θέλει να επενδύσει στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόσβαση στην χρηματοδότηση, πώς δεν είναι πρόβλημα. Μπορείτε να μας πείτε λεπτομέρειες. Και από ό,τι κατάλαβα, η αναλογία ανάμεσα στην παραγωγή ενέργειας και τα δίκτυα ηλεκτρισμού γέρνει προς τη μεριά της παραγωγής ενέργειας. Ωστόσο, οι επενδύσεις που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη των δικτύων είναι περίπου 60% των επενδύσεων ε, στην παραγωγή ε, ενέργειας. Ιδιαίτερα στον τομέα των ανανεώσιμων που είναι απαραίτητες. Είπατε και αναφέρετε και σε μία σας διαφάνεια ότι νέα χρηματοδοτικά μέσα και μοντέλα χρηματοδότησης, γιατί τελικά οι επενδύσεις αυτές στην ουσία πληρώνονται από τους πελάτες εν τέλει. Δεν έχει σημασία αν είναι ιδιωτικές ή εθνικές από τον προϋπολογισμό. το τέλος το κόστος είναι ψηλότερο και οι πελάτες πληρώνουν τα πάντα. Αλλά ποιος θα ξεκινήσει τις επενδύσεις? Θα είναι αποφάσεις ιδιωτών επενδυτών, εθνικών επενδυτών ή ίσως της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ποιο θα πρέπει να ξεκινήσει, μπορείτε εσεί να μας δώσετε κάποια ιδέα. Γιατί τελικά οι πελάτε θα πληρώσουμε, αλλά κάποιο πρέπει να κάνει την αρχή για να υλοποιηθούν όλα αυτά. Any Άλλο ζητάει το λόγο, όχι. Ωραία λοιπόν, να σας ζητήσω να μας απαντήσετε αγαπητοί ε, καλεσμένοι μας. Με την ίδια σειρά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 το ETS είναι πολύ καλή ερώτηση. Βέβαια ο στόχος της πρωτοβουλίας που μπορεί να αναλυφθεί στο πλαίσιο του ETS είναι να είναι ψηλότερη η τιμή και είναι μια σωστή παρέμβαση ώστε να δοθούν κίνητρα για επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές και στην μειχτή παραγωγή. Εάν αυξηθεί η τιμή του διοξιδίου του άνθρακα, του διοξιδίου του άνθρακα, τότε θα αυξηθεί και η τιμή του ηλεκτρισμού. Και τότε οι ανανεώσιμες θα γίνουν πιο επικερδείς και ανταγωνιστικές, χωρίς ε, ε, επιδοτήσεις. Από μακροοικονομική άποψη λοιπόν κερδίζει κανείς αν αυξήσει την τιμή του διοξιδίου του άνθρακα και πετυχαίνει και τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου. Ναι, μεταβλητό κόστος ε, του, ε, της περιθωριακού εργοστασίου. Ε, η τιμή τώρα είναι πολύ χαμηλή για να προσελκύσει επενδύσεις. Οι επενδύσεις ανανεώσιμες γίνονται μόνο με βάση τις επιδοτήσεις. Εάν καταργηθούν οι επιδοτήσεις δεν θα γίνουν πια ε, επενδύσεις στην παραγωγή ούτε για τις ανανεώσιμες ούτε για τις συμβατικές τεχνολογίες. Αυτό είναι κομμάτι της απάντησης λοιπόν. Και αν η τιμή του διοξιδίου φτάσει σε εντός εισαγωγικών λογικά επίπεδα, Ίσως να μην χρειάζεται μηχανισμός ε, αμοιβή της ε, παραγωγικής δυνατότητας. Θα μπορούσε δηλαδή με άλλα λόγια να ρυθμιστεί αυτό από την πλευρά της ε, παροχής. Όσον αφορά τις επενδύσεις σε δίκτυα, ο αντίκτυπος της αποκεντρωμένης παραγωγής, καταρχήν η αποκεντρωμένη παραγωγή εξετάζεται στις διάφορες υποθέσεις που χρησιμοποιήσαμε για να κάνουμε τη μελέτη μας και να σας παρουσιάσουμε αυτά τα στοιχεία. Όμως ε, φυσικά όλα αυτά εξαρτώνται και από την ε, εξέλιξη της τεχνολογίας. Αν για παράδειγμα οι συσσωρευτές, οι μπαταρίες είναι λύση, και αν γίνουν επενδύσεις σε αυτές, ας πούμε αναφέρθηκα στη Γερμανία όπου 30% των νέων εγκαταστάσεων είναι εξοπλισμένες με ε, στήλες ισόρευσης ε, εφεδρικές, τότε δεν ε, θα μιλήσουμε τόσο για ανάπτυξη δικτύων. Οι τεχνολογικές εξελίξεις όσον αφορά την αποθήκευση θα καθορίσουν και τις επενδύσεις που θα απαιτηθούν για τα δίκτυα και οι τιμές σύνδεσης, τα τέλη σύνδεσης μάλλον, θα επηρεάσουν και τις επενδύσεις σε δίκτυα. Θα πρέπει καταρχάς να εξελιχθούμε σε ένα δίκαιο τμήμα του κόστους ε, επενδύσεων στις, ε, στα δίκτυα ε, που θα επιβαρύνουν τους παραγωγούς, ώστε να έχουμε ένα βέλτιστο σύστημα κόστους που θα το ελαχιστοποιεί ταυτόχρονα το ίδιο το κόστος. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο σε αυτό το πλαίσιο. Ευελιξία και το μερίδιο της αποθήκευσης ώστε να υπάρχει δυνατότητα εξισορρόπησης των υπηρεσιών. Αυτό το μερίδιο και η συμβολή της αποθήκευσης θα εξαρτηθεί από πολλά πράγματα, όχι μόνο από την τεχνολογία, διότι γίνεται έρευνα αυτή τη στιγμή για νέες τεχνολογίες αποθήκευσης, χημική, και, χημική αποθήκευση κτλ. ή ε, ενέργεια σε ε, αέριο, υδρογόνο, ένα σωρό ανοιχτά ζητήματα από την άποψη της τεχνολογίας, αλλά Υπάρχουν και ζητήματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από τις αρχές, από τους πολιτικούς και αναφέρομαι στη ε, ε, τέλη για τα δίκτυα αλλά και για το ρυθμιστικό, ρυθμιστικό πλαίσιο. Για παράδειγμα η ιδιοκτησία είναι σημαντικό θέμα. Οι ε, φορείς που διαχειρίζονται τα δίκτυα θα μπορούν να διαχειρίζονται και την αποθήκευση. Αυτό δεν έχει ρυθμιστεί αλλά είναι πολύ σημαντικό για τους φορείς στην διαχείριση στο τομέα του ηλεκτρισμού. Επίσης, η δίκτυο και αποθήκευση. Θεωρείτε ότι η αποθήκευση είναι παραγωγός ή χρήστης. Ο, δηλαδή, θα χρεώσετε και την παραγωγή και την αποθήκευση. Μάλλον, ε, και την παραγωγή και τον χρήστη και τις ε, εγκαταστάσεις αποθήκευσης. Ορίζοντας λοιπόν το αριθμιστικό πλαίσιο σε σχέση με την ιδιοκτησία, θα ορίσετε και το ποσοστό ανάπτυξης της αποθήκευσης και το μερίδιο που μπορεί να προσφέρει η αποθήκευση στο νέο σύστημα. Σε σχέση με την ψηφιοποίηση είναι πάρα πολύ σημαντική και η συμμετοχή των πολιτών είναι μια φιλοδοξία του πακέτου του ναι, όντως να αυξηθεί η συμμετοχή των πολιτών. Αλλά και εκεί χρειάζονται διάφορα μέσα, όπως οι ευφυείς τιμές, οι δυναμικές τιμές, όπου ρυθμίζονται οι τιμές, τις ορίζουμε αλλά δεν μπορούμε έτσι να δώσουμε κίνητρα στους πολίτες ώστε να αποτελέσουν έναν ενεργό φορέα, έναν ενεργό παράγοντα στην ενεργειακή αγορά. Για το συγκεκριμένο τομέα χρειάζεται από τη μια πλευρά η τεχνολογία, ευφυή κουτιά, smart boxes, ευφυείς συσκευές, αλλά και κατάλληλες πολιτικές ταυτόχρονα παράλληλα. Αυτό είναι το που, αυτό που μας λένε τώρα για τη χρηματοδότηση οι ε, φορείς ε, ότι το κόστος της χρηματοδότησης δεν είναι πολύ μεγάλο ζήτημα. Το, η κερδοφορία είναι ζήτημα. Εάν μπορεί κανείς να εντοπίσει επικερδή project, έργα, ε, τότε δεν είναι πρόβλημα να βρει και συνεταίρους και να βρει τα λεφτά. Η κερδοφορία και ο κίνδυνος είναι τα θέματα. Δηλαδή, ρυθμιστικός κίνδυνος, ήδη αναφέρθηκα στο θέμα της ρύθμισης δύο-τρεις φορές, ρυθμιστικός κίνδυνος, βεβαιότητα για τους επενδυτές, σιγουριά και τεχνολογική κίνδυνη είναι επίσης αρκετά υψηλή και έπειτα έχουμε και τον οικονομικούς κινδύνους ποια θα είναι η τιμή και ποιο θα είναι το περιθώριο αύριο μεθαύριο, λαμβάνοντας υπόψη τις διάφορες ε, αβεβαιότητες που ε, οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε στον τομέα του ηλεκτρισμού. Και τέλος, Τέλος, σε σχέση με τις επενδύσεις, νομίζω θα πρέπει να δούμε τις ρυθμιστικές επενδύσεις και τις επενδύσεις στην ελεύθερη αγορά. Δηλαδή, οι διαχειριστέ των δικτύων θα πρέπει να κατευθύνονται με σαφείς στόχου και σαφείς κανόνε που ορίζουν οι αρχές. Ενώ οι επενδύσεις στην παραγωγή, αποθήκευση, εξοπλισμό από την πλευρά της ζήτησης. Ε, εκεί είναι ελεύθερη αγορά και εκεί θα πρέπει να ηγηθούν οι ιδιώτες επενδυτές όμως επί τη βάση ενός κατάλληλου και πρόσφορου ρυθμιστικού πλαισίου. Uh, Νομίζω, και αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, δεν είναι κάτι το οποίο συμπεριλάβαμε στην έκθεση, στο εφιστάμενο πλαίσιο δεν υπάρχει καμία άλλη εναλλακτική στο εφιστάμενο δηλαδή πλαίσιο και λαμβάνοντας υπόψη το ότι οι τιμές της αγορές χονδρικής επηρεάζονται μόνο από το κειμενόμενο κόστος, δεν υπάρχει καμία άλλη εναλλακτική. Επομένως χρειαζόμαστε ένα μηχανισμό αποζημίωσης των ικανοτήτων ηλεκτροπαραγωγής προκειμένου να μπορούμε να έχουμε το πετώμενο αυτό επίπεδο. Γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιούν αυτή την επιλογή πολλά κράτη-μέλη. Είναι μια προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή, η οποία όμως είναι αποδεκτή, διότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία ενιαία λύση η οποία είναι επαρκής και κατάλληλη για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, μια προσέγγιση από τη βάση προς τα πάνω μπορεί να αναποδεκτεί αρκεί να βασίζεται σε συγκεκριμένες ανάγκες των συγκεκριμένων κρατών μελών. Κάποια στιγμή όμως θα χρειαστεί και μια γενική ενιαία ευρωπαϊκή λύση, εκ των άνω προς τα κάτω, προκειμένου να έχουμε και ένα καλύτερο συντονισμό των πρωτοβουλειών και προκειμένου να ανοίξουμε τις αγορές των κρατών μελών, οι οποίες θα μπορούν πλέον, τα οποία κράτη-μέλη θα μπορούν να συμμετέχουν περισσότερο στις αγορές γειτονικών κρατών μελών. Τα όσα συμβαίνουν λοιπόν σήμερα δεν είναι μη αποδεκτά σε καμία περίπτωση, αλλά σιγά σιγά θα πρέπει να αρχίσουμε να κινούμεθα όλοι προς ένα κοινό στόχο, ο οποίος βέβαια θα πρέπει να είναι και από κοινού καθορισμένος. Η κυρία Γίεργουτ, να προσθέσω μόνο κάποια πράγματα, τα οποία ενδεχομένως να μην καλύψαμε, η έκθεση βασίζεται περισσότερο στο ευρωπαϊκό επίπεδο και στην αξιολόγηση του ευρωπαϊκού επίπεδου. Δεν έχουμε αριθμητικά δεδομένα για επιμέρου κράτη-μέλη για τα περισσότερα ζητήματα. Παρ' όλα αυτά, κάναμε μία εκτεταμένη αξιολόγηση κάποιων υφιστάμενων σεναρίων πολιτική και αν δείτε το παράρτημα τη έκθεση, μπορείτε να βρείτε εκεί πέρα περισσότερε λεπτομέρειε. Σε επίπεδο κράτου μέλου αυτή τη φορά. Νομίζω ότι όλα τα υπόλοιπα καλύφθηκαν από το συνάδελφο. Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Ήταν πραγματικά Πολύ ενδιαφέρουσε παρουσίαση αυτή και πάρα πολύ σημαντική για την Επιτροπή μας, προκειμένου να καταφέρουμε να συμβάλλουμε κι εμείς στην διαμόρφωση της ε, τοποθέτησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το χειμερινό νομοθετικό πακέτο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν για την παρουσίασή σας, καθώς επίσης και τις απαντήσεις που δώσετε σε ερωτήσεις των συναδέλφων. Αγαπητοί συνάδελφοι, ας περάσουμε τώρα στο σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης. Ορθώνει ο Πρόεδρο στο σημείο 4 τη ημερήσια διάταξη, προαγωγή τη ε, σύνδεση, τη συνδεσιμότητα μάλλον στο διαδίκτυο στι τοπικέ κοινότητε. Εισηγητή είναι ο κύριο Κάρλο Ζωρίνιο και όπω θα θυμάστε, το Σεπτέμβριο του 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε έναν κανονισμό με τίτλο «Προαγωγή της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες». Το πεδίο εφαρμογή τη πρόταση αυτή κανονισμού είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο. Συνδεσιμότητα σε δίκτυα σύρματα Wi-Fi για όλους τους πολίτες και για όλους τους επισκέπτες σε όλους τους δημόσιους χώρους παντού στην Ευρώπη μέσω της πρωτοβουλίας Wi-Fi for EU, ασύρματα δίκτυα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς είμαστε η καθήλυνα αρμόδια επιτροπή για την πρόταση αυτή, αλλά οι επιτροπές μεταφορών, η Επιτροπή Προπολογισμών και η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης είναι γνωμοδοτικές επιτροπές, σύμφωνα με το άρθρο 53 του κανονισμού μας. Η δική μας αρμοδιότητα και ευθύνη είναι ξεκάθαρη πάντως. Κύριε Ζωρίνιο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, Το σχέδιο της έκθεσης αυτής της σημαντικής πρωτοβουλίας Wi-Fi for EU ε, ασύρματη σύνδεση για την Ευρωπαϊκή Ένωση, προώθηση δηλαδή της συνδεσιμότητας των τοπικών ε, ε, αρχών είναι, δείχνει μάλλον σαφώς και τονίζει ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να συνδεθούμε συνδεθούν μάλλον οι Ευρωπαίοι πολίτες με τους θεσμούς και με το ευρωπαϊκό όραμα. Και στην ε, περίπτωση της ε, ψηφιακής ένωσης, αυτό σημαίνει πως οι πολίτες θα πρέπει να κατανοήσουν και να διαπιστώσουν με τα ίδια τους τα μάτια τα πλεονεκτήματα που μπορεί να φέρει η ψηφιακή ενιαία αγορά στην καθημερινή του ζωή. Είναι σημαντικό λοιπόν αυτό να συνοδεύεται από ένα, ένα πλαίσιο της τεχνολογικής εξέλιξης που επηρεάζει τη φύση της οικονομίας αλλά και της κοινωνίας μας. Αυτή η πρωτοβουλία έχει ακριβώς αυτό το στόχο να δώσει, να προσφέρει στους πολίτες συγκεκριμένα ωφέλη και ταυτόχρονα να λειτουργήσει ως ένα πρόγραμμα δοκιμαστικό και ένα υπόδειγμα του πώς θα θέλαμε να εξελιχθεί μια ε, ε, ευρωπαϊκή κοινωνία Gigabyte που να περιλαμβάνει όλους, να είναι καθολική, ενώ ταυτόχρονα θα είναι και πρωτοπόρος ε, τεχνολογικά σε αυτό το αναθεωρημένο σχέδιο, το οποίο συνέταξα αφού ήρθα σε επαφή με τους θεσμούς, ήρθα και μάλιστα στην ε, Περιφερειακή Επιτροπή όταν, την ημέρα μάλιστα που ενέκριναν τη δική τους ε, γνωμοδότηση, άκουσα τους διάφορους ε, φορείς, παρόχους, ακτιβιστές, καθώς και τους κοιόδης μας εισηγητές φυσικά που συνέβαλαν πολύ σημαντικά και μάλιστα έγιναν και δύο δημόσιες Ακροάσει ε, από την Επιτροπή μας στο πλαίσιο του πακέτου των τηλεπικοινωνιών, Telecom. Με βάση αυτά λοιπόν η έκθεσή μου περιλαμβάνει φυσικά διάφορες ιδέες, αλλά πέντε βασικά θέματα είναι αυτά που θέλω να τονίσω. Πρώτο, εστιάζουμε στην ποιότητα της εμπειρίας. Πρέπει να εγγυηθούμε την ουδετερότητα του ε, δικτύου, την ουδετερότητα την τεχνολογική, την ουδετερότητα, την οικονομική, δηλαδή κανένας να με μένει εκτός επειδή δεν μπορεί να πληρώσει, να εγγυηθούμε την γεωγραφική ουδετερότητα, κανείς να με μένει εκτός επειδή κατοικεί μακριά ε, ή πάνω σε κάνα βουνό ή σε κάποιο μέρος απομακρυσμένο από το κέντρο, αλλά ε, ε, υπάρχει και ένα στοιχείο που δεν μπορούμε να είμαστε ουδέτεροι, δηλαδή η η ποιότητα αυτής της εμπειρίας θα πρέπει να είναι υψηλή. Και αυτός είναι ο μόνος τρόπος όπου θα μπορέσουμε να εγγυηθούμε την αντοχή αυτού του project στην εξέλιξη των τεχνολογιών χωρίς αυτό να πλήξει την ουδετερότητα. Γιατί οι τεχνολογίες θα εξελιχθούν κι άλλο. Αλλά θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι ώστε κάθε φορά η εμπειρία αυτή να είναι της ποιότητας. Επίσης υπάρχει αρχή της ε, μοναδικής ταυτοποίησης, ε, ε, one login only. Τρίτον, απλότητα των διαδικασιών και αυτό είναι λογικό γιατί θέλουμε να είναι απλό, γρήγορο και αποτελεσματικό. Και γι' αυτό και έχουμε την ιδέα της χρηματοδότησης με voucher ή κριτήρια της σειράς άφηξης, ούτως ώστε κάθε χώρα αυτό είναι στην πρόταση τη Κομισιόν, όχι στη δική μου έκθεση. Δηλαδή, λέει και ο πρώτο που έρχεται, ο πρώτο θα εξυπηρετείται. Εμεί λέμε ναι, ότι ο πρώτο που φτάνει θα πρέπει να εξυπηρετείται, αλλά κάθε χώρα μπορεί να εκπονήσει το δικό τη πρόγραμμα εργασία με συγκεκριμένε προτεραιότητες. Κάποιοι μπορεί να δώσουν προτεραιότητα, α πούμε, στι ε, ζώνε τη υπαίθρου, άλλοι στα αστικά κέντρα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θα πρέπει να είναι εγγυημένο είναι η συνοχή και η συνιστόσα τη καθολικότητα. Επίσης, ε, δεν μας ε, πειράζει, δεν, δεν, δεν, δεν είναι σημαντική τόσο αν είναι ιδιωτική ή, ε, ή κρατική ή επένδυση. Θα προέπει ωστόσο να γίνουν αυτά εντό σύντομου χρονικού διαστήματος με χρηματοδότηση τόσο δημόσια όσο και ιδιωτική, ώστε να εγγυηθούμε πως αυτά τα project θα αναπτυχθούν και θα υλοποιηθούν επί τόπου. Ε, Κύριε Πρόεδρε, θα μας πει έχουμε, ε, είναι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών. Ε, θέλω να προτρέξω και πρέπει να πω ότι πέρα από ενδεχόμενε τροπολογίες που μπορεί να καταθέσουν οι συνάδελφοι, να ευχαριστήσω την εξαιρετική συνεργασία που είχα με όλους τους κοιόδης και έχω την πρόθεση να ε, καταθέσω και εγώ δύο τροπολογίες ε, που αποσαφηνίζουν την αναφορά στο απλοποιημένο μοντέλο για τον έλεγχο της χρήσης των χρημάτων που θα χρησιμοποιηθούν, που πρέπει να είναι απλοποιημένο, πρέπει να είναι και αυτό απλοποιημένο και ε, γρήγορο. Και από την άλλη πλευρά μια άλλη τροπολογία που αποσαφηνίζει τους περιορισμούς, γιατί αυτό το project έχουν να κάνουν με τη ταχύτητα, με τον όγκο, με τη δυνατότητα πρόσβασης και Όπως όλα τα προγράμματα, τα ψηφιακά, έτσι και εδώ θα υπάρξουν κάποιοι συγκεκριμένοι τεχνικοί περιορισμοί. Το project αυτό, τελειώνω πρόεδρε, είναι ένα project όχι πολύ μεγάλο από άποψη επενδύσεων, αλλά είναι πολύ συμβολικό και είναι πολύ σημαντικός και ο χρονισμός αυτού του project να γίνει γρήγορα, να ξεκινήσει γρήγορα. Είναι δυνατόν να ξεκινήσει ήδη από το επόμενο εξάμεινο αυτό για να σηματοδοτήσει ε, ολόκληρο το ψηφιακό πακέτο. Θα πρέπει να γίνει δηλαδή αυτό το πακέτο να εφαρμοστεί τώρα. Είναι ένα καλό ε, και απλό πρόγραμμα τώρα είναι πολύ πιο σημαντικό από ένα περίπλοκο και πιο μεγάλο πρόγραμμα του χρόνου. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Σιγητά. Και τώρα, εξ του ΕΛΚ, η κυρία Αν Σάντερ. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Εγώ θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή Κάρλο Ζωγίνιο για το σχέδιο έκθεσης που επιτρέπει να αποσαφηνίσουμε κάποια σημεία του κανονισμού. Για να σα θυμίσω, αυτό το πρόγραμμα επιτρέπει τη χρηματοδότηση με 20.000 ευρώ τοπικέ αρχέ που θέλουν να εγκαταστήσουν ε, ε, δυνατότητα Wi-Fi στους δημόσιους χώρους και να προσφέρουν δωρεάν σύνδεση στους συμπολίτες τους. Όπως έλεγαμε και την περασμένη φορά, η πολιτική μου ομάδα υποστηρίζει αυτή την πρόταση, γιατί οι πολίτες χρειάζονται μια Ευρώπη που να είναι χρήσιμη, συγκεκριμένη, απτή ε, και που να είναι πραγματικά ορατή στην καθημερινή ζωή τους. Ωστόσο, θα πρέπει να διευκρινίσουμε κάποιες πτυχές. Η μία είναι να μην δημιουργήσουμε φρούδες ελπίδες. Το πρόγραμμα αυτό έχει μόνο στη διαθεσία του 120 εκατομμύρια ευρώ. Από τις 90.000 λοιπόν δήμους της Ευρώπης, μόνο 8 με 10.000 θα μπορέσουν να το χρησιμοποιήσουν. Αυτό το πρόγραμμα θα πρέπει να μπορέσει να συμπληρωθεί από άλλες πηγές χρηματοδότηση, όπως για παράδειγμα τα όσα απομένουν από τα διαρθωτικά ταμεία. Είμαι υπέρ λοιπόν της τροπολογίας 18 του σχεδίου έκθεσης. Στη συνέχεια, το σχέδιο κανονισμού προβλέπει μόνο η συνδεσιμότητα υψηλή ταχύτητα να είναι επιλέξιμη, Όμω, όπω θυμίζει και ο ίδιο ο εισηγητή στην τροπολογία του υπαρθμών 7, τα τρία τέταρτα των ευρωπαϊκών σπιτιών στι περιοχέ τη Υπέθρου δεν έχουν σταθερό γρήγορο ίντερνετ. Γι' αυτό θα πρέπει να μειωθούν αυτέ οι απαιτήσει για πολύ μεγάλη ταχύτητα, ώστε τα προγράμματα αυτά να χρησιμοποιηθούν σε ζώνε όπου πραγματικά υπάρχει ανάγκη με υπέρ λοιπόν της ιδέας της τροπολογίας 14. Τέλος, είμαι υπέρ της ιδέας ενός συστήματος μοναδικής ταυτοποίησης που θα ισχύει για όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως προβλέπεται στην τροπολογία 3. Αντίθετα, δεν συμμερίζομαι την άποψη του του εισηγητή για την απαγόρευση κάθε περιορισμού συμπεριλαμβανομένου ε, του θέματος του όγκου ή του χρόνου. Θα πρέπει να μπορούν οι τοπικές αρχές να προλάβουν τις ε, καταχρήσεις και να περιορίσουν την πρόσβαση σε site των οποίων το περιεχόμενο είναι παράνομο. Επίσης ε, πρέπει και οι δήμοι να είναι επιλέξιμοι, ώστε να, ε, μάλλον ομάδες δήμων να μπορούν να είναι επιλέξιμες ώστε να διευκολυνθεί το εγχείρημα αυτό. Πιστεύω εν τέλει πως έχουμε τους ίδιους στόχους και ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα ώστε να μπορέσουν να γίνουν οι πρώτες επιλογές ε, πριν το τέλος του καλοκαιριού. Επιμένω δε ότι πρόκειται για ένα project που μπορεί να επιτρέψει να φανεί μια Ευρώπη συγκεκριμένη, ρεαλιστική, κοντά στους πολίτες και δεδομένου του γενικού ε, της γενικής ατμόσφαιρας που επικρατεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πιστεύω πως είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το σημείο. Ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφε Τελίτσκα για την ομάδα των Φιλελευθέρων. Ευχαριστώ Πρόεδρε, συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. να πω ότι εκτιμώ ιδιαίτερα την ε, στάση του εισηγητή. Ήταν χαρά που συνεργαστήκαμε εδώ. Βλέπουμε ότι σε κάποια κράτη-μέλη ακόμα δεν έχουμε την ψηφιακή κουλτούρα, θα λέγαμε, που να δείχνει προφανώς ότι κάθε δήμος, κάθε κοινότητα με κάποιο τρόπο έχει σύνδεση με Wi-Fi. Εδώ χρειάζονται εθνικές επενδύσεις και αυτό το πρόγραμμα. Προφανώς ε, αυτά που συζητάμε δεν θα αλλάξουν άρδιν την κατάσταση γιατί τα, οι πόροι είναι περιορισμένοι. Θα προσέθετα άλλωστε ότι δεν είναι δουλειά της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υποκαταστήσει τη χρηματοδότηση ε, από τους εθνικούς ή ε, τοπικούς προϋπολογισμούς. Αυτό που είναι εποφελές και χάρηκα γιατί είχαμε επικοδομητική συνεργασία που και αμοιβαία αποδεκτό αποτέλεσμα ότι θα δώσει μια δυναμική. Θα επιταχυνθούν οι αλλαγές στα κράτη-μέλη, κυρίως στα κράτη-μέλη όπου αυτή η κουλτούρα η ψηφιακή δεν έχει οριμάσει. Και βέβαια υπάρχουν διάφοροι δήμοι, διάφοροι δικαιούχοι από μακρισμένες περιοχές κλπ. Τα έχουμε πει αυτά και στο παρελθόν. Τώρα, για το σχέδιο πρότασης. Είναι καλό σχέδιο. Αντικατοπτρίζει και τις συζητήσεις που προηγήθηκαν. Υπάρχουν και κάποια θέματα που μένουν να εξεταστούν. Και εκεί μπορεί να καταθέσω εμπροθέσμες τροπολογίες. Σημαντικό είναι να, ε, ότι έχουμε ένα σύντομο πρόγραμμα εδώ που δεν θα συνεχιστεί, αλλά που θα έχει έναν αντίκτυπο που θα κάνει τη διαφορά. Κατόπιν τούτου πρέπει να πούμε ότι το πώς θα ε, αλληλεπιδράσει η Κομισιόν ε, με τους ενδιαφερόμενους θα συμβάλλει στην αλλαγή της κουλτούρας και θα έχουμε και παρεπόμενα έμεσα ωφέλη. Επίσης υπάρχει και αυτό το θέμα του συνδυασμού ενδεχομένως αυτού του προγράμματος με άλλα χρηματοδοτικά μέσα και διαρθρωτικά ταμεία. Μπορεί αυτό να το βλέπω λίγο διαφορετικά από τη στην τροπολογία 18 που δεν ξέρω τι σημαίνει ανάπτυξη συμπληρωματικών υπηρεσιών. Αν το θέμα είναι η συμπληρωματικότητα, συμφωνώ όμως. Γιατί θέλουμε να έχουμε πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα και με τους περιορισμένους πόρους. Η γεωγραφική ισορροπία αναφέρθηκε. Ο κύριος Σωρίνιο νομίζω βρήκε τη σωστή ισορροπία εδώ με την ε, τροπολογία του. Ε, είναι θεμητή η τροπολογία. Επίσης, κοιτάξαμε και το θέμα πιθανής στρέβλωσης του ανταγωνισμού. Ε, θα θυμάστε ότι ε, εγώ έθεσα το θέμα. Ε, είχα πει ότι θα υπάρχει κάποια παρεμβολή μεταξύ των δικαιούχων αυτού του προγράμματος του καινούριου και κάποιων άλλων σε, στους ε, Δήμους όπου θα αναπτυχθεί το πρόγραμμα. Αυτό θα πρέπει τουλάχιστον στις αιτιολογικές σκέψεις να το πούμε. Την Κομισιόν κατά την εφαρμογή θα πρέπει να αποφύγει καταστάσεις που μπορεί να ε, επηρεάσουν, ίσως όχι πολύ, αλλά μπορεί να δημιουργήσουν ένα ε, δυσμενές περιβάλλον. Να δούμε λίγο και την τροπολογία 11 προαγωγή της καθολικής πρόσβασης ε, των πολιτών στα ωφέλη της κοινωνίας των πληροφοριών. Θα πρέπει να το σκεφτούμε λίγο αυτό για να δούμε πώς θα συνάδει αυτό και με το θέμα των καθολικών υπηρεσιών καθ' αυτών. Γενικά θα έλεγα κυρία Πρόεδρε, κυρία Ζουρίνιο, Ζουρίνιο κυρία συνάδελφοι, ότι θα καταθέσω κάποιες τροπολογίες που δεν θα αλλάξουν όμως στις βασικές γραμμές το σχέδιο που θεωρώ ότι είναι καλό. Το πιο σημαντικό είναι να το αναπτύξουμε και να το εφαρμόσουμε το ταχύτερο δυνατόν, να έχουμε την πρώτη, τις πρώτες προσφορές, ε, την εκδήλωση ενδιαφέροντος και να φροντίσουμε να έχουμε καλό feedback από τους παρέχοντες της υπηρεσίες. Είναι πολύ σημαντικό και να, ε, από εκεί θα ξεκινήσουμε. Ευχαριστώ. κύριος Ηλικιώτης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συναδελφό τον Κάρλο Ζωρινίου για την παραγωγική συζήτηση που είχαμε στην πρώτη συνάντηση των σκιωδών εισηγητών και για ιδιαίτερα για τη θέση που ανάπτυξε όσον αφορά την προαγωγή τη σύνδεση στο διαδίκτυο στι τοπικέ κοινότητε. Εμεί συμφωνούμε με τη θέση του εισηγητή πω πρέπει να στηρίζουμε αυτή την πρωτοβουλία ώστε να υπάρχει δωρεάν ασύρματη συνδεσιμότητα σε χώρου όπου παρέχονται δημόσιε υπηρεσίε, όπως οι δημόσιες διοικήσεις, οι βιβλιοθήκες, τα νοσοκομεία. Ωστόσο, θεωρούμε σημαντικό να αναπτυχθεί η πρόταση ώστε να καλύπτει τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, χώρους δημόσιων συγκοινωνιών, καθώς και άλλους χώρους της κοινωνικής ζωής. Επίσης, συμφωνούμε απόλυτα με τον εισηγητή ότι είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί πως ο διαθέσιμος προορισμό θα κατανεμηθεί με γεωγραφικά ισορροπημένο τρόπο. Για την ομάδα μα είναι προτεραιότητα να επιφορηθούν από την ασύρματη συνδεσιμότητα ιδιαίτερα τα κράτη και οι περιοχέ που είναι λιγότερο ανεπτυγμένε, τα νησιά και οι ορεινέ περιοχέ, οι παραμεθόριε, οι απομακρυσμένε και οι πρόσιτε περιοχέ. Στόχο μα βέβαια είναι να και ανάγκε όλων των πολιτών, να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό δημόσιο όφελο και να δοθεί δυνατότητα στου πολίτε από όλα τα κοινωνικά στρώματα να αποφεληθούν από τα πλεονεκτήματα τη Όμω θα ήθελα να σημειώσω επίση ότι θα καταψηφίσουμε την πρόταση τη Κομισιόν, η οποία υποστηρίζει πω ο προπολογισμό θα κατατίθεται κατά κανόνα με βάση σειρά παραλαβή των προτάσεων. First come, first serve. Ε, αντί αυτού, τονίζουμε πω πρέπει να ενημερωθούν άμεσα τα κράτη και οι τοπικέ αρχέ σχετικά με τη σχεδιαζόμενη δράση και του σχετικού όρου, αλλά και να στηριχτούν επαρκώ ώστε να ξεκινήσουν άμεσα τις προεργασίες για την υποβολή αιτήσεων. Εξίσου σημαντικό είναι να μην παραγνωριστεί η σημαντικότητα της συμμετοχής μελών των τοπικών κοινοτήτων στην υλοποίηση της όποιας δράσης. Δηλαδή στο καθορισμό των κέντρων του δημόσιου βίου όπου θα υπάρξει εγκατάσταση δωρεά σημείων ασύρματης πρόσβασης διασφαλίζοντας έτσι τη μεγαλύτερη προσθέμενη αξία για την κοινότητα. Τέλος, θα πρέπει να διασφαλίσουμε πως η τοπική ασύρματη συνδεσιμότητα θα πρέπει να λογίζεται ω δωρεάν μόνο εφόσον παρέχεται χωρί χρέωση. Είτε αυτή γίνεται υπό μορφή άμεση πληρωμή, είτε έναντι άλλου τμήματο, συμπεριλαμβανομένη μεταξύ άλλων τη διαφήμιση και τη παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Και προ αυτή την κατεύθυνση θα είναι και οι τροπολογίε που, ε, που θα καταθέσουμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. πολύ, Πρόεδρε. Προσεγγίζουμε με αυτή την έκθεση την ουσία της ε, συνδεσιμότητας ε, των πολιτών στις τοπικές ε, περιοχές, μιλώντας για το Wi-Fi ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά στις ζώνες της Υπέθρου, όπως και στη δική μου περιφέρεια, από την οποία προέρχομαι, δηλαδή τη Γαλλικία. Θέλω να ευχαριστήσω τον Κάρλες για αυτή την εξαιρετική του πρόταση, γιατί δίνει, ε, έχει πραγματικά χτυπήσει στο κέριο σημείο, μιλώντας για σημεία πρόσβασης ε, και για χρηματοδότηση, μάλλον για, και προτείνοντας ένα σύστημα με μία μοναδική ταυτοποίηση, καθώς και το ότι η πρόταση ε, ε, η πρόσβαση να είναι ε, απεριόριστη, χωρίς κανέναν δηλαδή περιορισμό και επίσης ότι μιλά για τις λιγότερο ψηφιοποιημένες περιοχές. Το Ε, πιστεύω πως ε, η πρικοδότηση για αυτό το πρόγραμμα είναι πολύ μικρή και γι' αυτό θα πρέπει να περιλάβουμε εδώ και μια υποχρέωση υπηρεσίας, καθολικής υπηρεσίας, ώστε να εγγυηθούμε να μην, ότι δεν θα υπάρχει στο μέλλον ε, χρήση εμπορική αυτής της δομής που θα αναπτυχθεί με αυτά τα χρήματα. Αυτές είναι, αυτοί είναι οι προβληματισμοί μου, τους οποίους θα αναφέρω και στις τροπολογίες τις οποίες θα καταθέσω. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, συνάδελφε. Προθεσμία για τις τροπολογίες είναι η 5η, 2 Μαρτίου. Και τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τη Γενική Διεύθυνση Connect που εκπροσωπείται από τον επικεφαλής ε, της μονάδας, τον κύριο Ντιπουή. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή και τους σκιώδες για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Χαιρετίζουμε ιδιαίτερα τις θέσεις που εκφράστηκαν σήμερα και αυτές που υπάρχουν στην έκθεση και πάνε προς την ίδια κατεύθυνση, όπως είδαμε στη διαδικασία του Συμβουλίου. Επίσης, σημεριζόμεθα εν πολλής την άποψη ότι είναι πολύ επίκαιρη η πρωτοβουλία που χρειάζεται πολύ τώρα και όσο ταχύτερα ε, συσταθεί και ε, εφαρμοστεί προς όφελος των πολιτών, τόσο το καλύτερο. Επίσης, χαιρετίζουμε το γεγονός ότι περισσότερες τροπολογίες είναι σημαντικές βελτιώσεις στο κείμενο, ε, τις αναφορές στο gigabit, ε, το ενιαίο σύστημα ταυτοποίησης, σύνδεσης, το γεγονός ότι θα είναι δωρεάν συνδεσιμότητα, οι αναφορές σε περισσότερους δημόσιους χώρους όπως χώρους πολιτισμού. Όλα αυτά συνιστούν σημαντικές βελτιώσεις στην αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα, σε ό,τι αφορά κάποια άλλα θέματα, εκεί έχουμε ορισμένε επιφυλάξεις. Ε, παρακολουθούμε τη συζήτηση για την ε, γεωγραφικά ισορροπημένη κατανομή, ε, τα, την αρχή το, του first come, first served. οι δύο αρχές δεν είναι ασυμβίβαστες μεταξύ τους. Αντίθετα υπάρχουν τρόποι να αντιμετωπίσουμε τα ειδικότερα αυτά χαρακτηριστικά και θέλουμε αυτά τα χαρακτηριστικά να τα δούμε σε επίπεδο προγράμματος εργασίας για να κάνουμε τις απαραίτητες τροπολογίες, προσαρμογές των διαφόρων κριτηρίων ε, ανάλογα με την αξιολόγηση κάθε ε, προσφοράς, ούτως ώστε η κατάσταση να αξιολογείται αναπερίπτωση ε, σε κάθε προκήρυξη. Αυτό είναι ένα κομμάτι μιας νεωτεριστικής προσέγγισης αυτής της πρωτοβουλίας. Θέλουμε πάρα πολύ το σύστημα αυτό να εφαρμόζεται τόσο εύκολα, ώστε κάθε κοινότητα οπουδήποτε στην Ευρώπη να μπορεί να το λειτουργεί ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όπως και μια άλλη κοινότητα πολύ πιο ανεπτυγμένη. Και παράλληλα θα είναι και ένα πρόγραμμα πολύ καινοτόμο. Δύο ακόμα παρατηρήσεις σχετικά με τις διαστάσεις της ουδετερότητας της τεχνολογίας είναι καταρχήν σημαντικό να υπάρχουν ξεκάθαρα σημεία πρόσβασης, συνδεσιμότητα, Wi-Fi θα είναι το βασικό σύστημα ε, που θα παρέχεται στους πολίτες. Αυτό δεν σημαίνει ότι ε, θα προσκρούσουμε στην ε, αρχή της ε, ουδετερότητα της σύνδεσης. Ε, αυτό θα εξακολουθήσει να ισχύει. Επίσης, η ουδετερότητα και οι διάφορες αναφορές στο ότι η συνδεσιμότητα θα πρέπει να μην υπόκειται σε κανένα περιορισμό. Ε, πιστεύουμε ότι εκεί μπορούμε να μπούμε σε μια άλλη συζήτηση που ίσως θα πρέπει να γίνει σε διαφορετικές διαπραγματεύσεις, όχι εδώ. Δηλαδή η πολύ υπερβολική κανονιστική προσέγγιση ενδεχομένως θα δυσχεράνει την εφαρμογή και την οριστικοποίηση του συστήματος και την ε, τελική νομοθεσία ε, σε, συνεργασία με το Συμβούλιο. Γι' αυτούς τους λόγους πιστεύουμε ότι θα πρέπει να διατηρήσουμε μια ευέλικτη στάση στην νομοθεσία και η καθαυτό διαχείριση αυτών των σημείων πρόσβασης να βρίσκονται στο κατάλληλο επίπεδο, σύμφωνα με την επικουρικότητα, δηλαδή μεταξύ των κοινοτήτων και των τοπικών παρόχων ε, διαδικτύου. καλό θα ήταν να υπάρχει συνένεση ε, εδώ στο Κοινοβούλιο και βεβαίως ε, ευχόμαστε γρήγορα να τελειώσουν οι διαδικασίες σας. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις παρατηρήσεις σας. Ακούσουμε τώρα πάλι τον ε, εισηγητή μας, τον κύριο Ζωρίνη, ο οποίος μπορεί να συνοψίσει κάπως τα συμπεράσματά του. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τους συναδέλφους συν εισηγητές, τον κύριο Σιλικιώτη, την κυρία το τον συνάδελφο Μπλανκολόπη, στην Επιτροπή, όλου όσοι πήραν το λόγο. Όντως θέλουμε να αναπτύξουμε μια κοινή, ένα κοινό όραμα. Γνωρίζουμε ακριβώς τι θέλουμε και γνωρίζουμε ποια είναι τα εμπόδια που θα πρέπει από κοινού να ξεπεράσουμε ώστε να βελτιώσουμε όλες τις τροπολογίες, ε, με, με όλες μάλλον τις τροπολογίες ε, που είναι πρόσδεκτες. Ε, είναι σημαντικό λοιπόν η έκθεση αυτή να απολοποιεί αλλά και να ελέγχει κάποια πράγματα ε, είναι σημαντικό και είναι και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού ε, Κοινοβουλίου είναι αυτός, ότι ορισμένα πράγματα να είναι μέσα σε αυτή την έκθεση. Γι' αυτό πρέπει να δούμε, όπως είπε και η συνάδελφος Σάντερ, πρέπει να, να, να επιμείνουμε περισσότερο στο θέμα των περιορισμών και το ζήτημα αυτών των περιορισμών να καθορίζεται. Επίσης, Έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο όσον αφορά το θέμα του ότι ο πρώτος που θα φτάσει να είναι και αυτός που θα εξυπηρετηθεί. Δεν συμφωνούσα και εγώ με αυτήν την ιδέα, όπω και ο συνάδελφο Μπλανκολόπης, αλλά με βάση αυτή την ιδέα, αν αυτή τη συνδέσουμε με τα προγράμματα εργασίας των εθνικών κρατών, μπορέσουμε, μπορούμε μάλλον να δώσουμε μια απάντηση απόλυτης επικουρικότητας. Δηλαδή τα όσα πρέπει να γίνουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο να γίνουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τα όσα μπορούν να γίνουν σε τοπικό να γίνουν σε τοπικό. Έχουμε δηλαδή κατά κάποιο τρόπο το ότι ο πρώτος που θα φτάσει θα είναι ο πρώτος που θα εξυπηρετηθεί, αλλά που ορίζεται από τις συγκεκριμένες συνθήκες που επικρατούν σε κάθε κράτος. Ναι, αυτό περιπλέκει κάπως τα πράγματα για την Κομισιόν, όχι όμως για το ίδιο το πρόγραμμα, δεν το καθυστερεί και βελτιώνει το τελικό αποτέλεσμα. Όπως για παράδειγμα το θέμα του προπολογισμού. Είναι σαφές ότι έχουμε 120 εκατομμύρια τα 70 είναι εγγυημένα από ό,τι ξέρω, τα 50 ακόμα όχι. Ε, αλλά ε, δυστυχώς, όπως είπε και ο συνάδελφος ε, Τελίτσα, ε, αυτά τα χρήματα θα πρέπει να συμπληρωθούν με ίδιους πόρους, με άλλου είδους στήριξη, ώστε τα project αυτά να πολλαπλασιαστούν και να διατηρηθούν, αλλά και έτσι ώστε όπως είπε ο συνάδελφος Μπλανκολόπες, να μπορέσουμε να φτάσουμε και να το ξεκινήσουμε ήδη από φέτος από τις τοπικές αρχές, αλλά να δούμε και αν μπορούμε να το επεκτείνουμε. Να, στον τομέα της παιδείας, της υγείας, του πολιτισμού. Δηλαδή, το project αυτό δημιουργεί πολύ ενδιαφέρουσες δυναμικές. Φανταστείτε, για παράδειγμα, μια τοπική αρχή που μπορεί να στηρίξει τι διάφορες οργανισμούς στην περιοχή. Ενώ και φανταστείτε ότι με τον προϋπολογισμό που έχουμε μόνο 10 μπορεί να χρηματοδοτηθούν από, τις, από αυτούς που ζήτησαν. Όμως αν δημιουργήσουμε με μεγάλη δυναμική με ένα σπουδαίο στόχο ε, να δούμε Πώς δηλαδή θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια δυναμική ώστε να επεκταθεί και να ανθίσει αυτό το πρόγραμμα. Ευχαριστώ και πάλι λοιπόν. Θα δεχτώ τι τροπολογίε σα, θα δούμε πώ μπορούμε να τι συνδυάσουμε ώστε να έχουμε ένα όσο γίνεται καλύτερο project για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Εμείς ευχαριστούμε κύριε Ζωρίνιο. Η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών είναι η 5η Δευτέρα Μαρτίου 2017 προφανώς. 12 το μεσημέρι. Επαναλαμβάνω, 2 Μαρτίου, 5η 2 Μαρτίου, 12 το μεσημέρι. Σας ευχαριστώ πολύ. Ας περάσουμε στο σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης, δημοσιονομικοί κανόνες που εφαρμόζονται στο Γενικό Προπολογισμό της Ένωσης. MMMFF Omnibus είναι ο τίτλος του κανονισμού αυτού. Πρόκειται για ένα συγκεκριμένο κανονισμό, έκτακτο κανονισμό, Υποσχέθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να επαναληφθεί τέτοια πρόταση κανονισμού κατά αυτόν τον τρόπο στο μέλλον δηλαδή να έχουμε έναν κανονισμό όμνιμπους για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, αλλά ότι θα έχουμε ξεχωριστές ε, προτάσεις για κάθε ξεχωριστό τομέα δαπανών. Ο δημοσιονομικός λοιπόν κανονισμός καθορίζει τις αρχές και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν για την κατάρτιση και την εκτέλεση του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τον έλεγχο των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την προτινόμενη αυτή αναθόρηση, η Επιτροπή στοχεύει να επιτύχει, να επιτύχει απλούστερους και πιο ευέλικτους κανόνες που θα πρέπει να βοηθήσουν στη βελτιστοποίηση των δαπανών και της επίδρασης του τρέχοντος πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου μέχρι το 2020. Η αναθεώρηση λοιπόν περιλαμβάνει εκτεταμένες αλλαγές, καταρχάς στους γενικούς δημοσιονομικούς κανόνες, το πρώτο μέρος της πρότασης δηλαδή, αλλά και αντίστοιχες αλλαγές στους κανόνες για τα τομεακά ταμεία και αλλάζει επίσης μια σειρά από ειδικέ διατάξεις στις ε, βασικές πράξεις των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκή ενωση και αυτό είναι το δεύτερο τμήμα της πρότασης κανονισμού. Αυτά είναι τα δύο σημαντικότερα τμήματα λοιπόν της προτινόμενου, του προτινόμενου κανονισμού. Όσον αφορά τώρα τις προτινόμενες τροποποίησεις όπου η ΙΤΡΑ έχει αποκλειστική αρμοδιότητα, οι, προτινόμενες, ε, οι προτινόμενες αλλαγές τροποποιούν ουσιαστικά τη διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη, τον κανονισμό κατευθυντηρίων γραμμών για τις τηλεπικοινωνίες, καθώς επίσης και το πλαίσιο στήριξης SST για την ε, παρακολούθηση και την επιτήρηση του διαστήματος. Πρόκειται για ένα ειδικό πλαίσιο στήριξης όσον αφορά το διάστημα παρακολούθηση και επιτήρηση του διαστήματο SST. Εν γέννη, οι αλλαγές αυτές όσον αφορά τις αποκλειστικές αρμοδιότητες Επιτροπής μας είναι περιορισμένες και τεχνικής θα έλεγα Αυτό είναι το σημαντικότερο συμπέρασμα, το πρωταρχικό συμπέρασμα στο οποίο καταλήγω. Οι υπηρεσίε Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Γενική Διεύθυνση Budget, Energy, Connect, Move, μα δώσανε λεπτομερεί εξηγήσει εδώ σε εμά, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τι ε, οποίε ε, έχουμε λάβει και στην έκθεση, στην επεξηγηματική δηλαδή έκθεση, στην οποία προσπαθώ να σας δώσω περισσότερες πληροφορίες, τις οποίες θεωρώ πιστικές. Πρόκειται για τις πληροφορίες που μας έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προφανώς όμως στη διάθεσή σας για τυχόν ανησυχίες ή ερωτηματικά που μπορείτε να έχετε. Είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να προετοιμάσουμε σωστά τη δική μας την τοποθέτηση. Όσον αφορά τώρα τις προτινόμενες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλαγές στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, δηλαδή για το CF και για τις κατευθύνες γραμμές στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, θα ήθελα εν προκειμένου να τονίσω το εξή ότι θα πρέπει οι αλλαγές αυτές να συντονιστούν με την πρόταση Wi-Fi for All, την οποία πρώτος, όπως ξέρετε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επεξεργάζεται εκ παραλλήλου, όπως άλλωστε είδαμε και σήμερα στο σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης. Μόλις τώρα συζητήσαμε την πρόταση αυτή Wi-Fi for All. Μην ξεχνάτε λοιπόν ότι Παράλληλα με την πρόταση αυτή κανονισμού θα πρέπει να εξετάζουμε και την πρόταση Wi-Fi for All και απευθύνουμε και στον Συγγετή κύριο Ζωρίνιο για λόγους εσωτερικής ε, συνέπειας όσον αφορά την ε, τοποθέτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε το ζήτημα των συνδυαστικών μηχανισμών blending facilities στα πλαίσια του CEF της διευκόλυνσης συνδέοντας την Ευρώπη στις συζητήσει που γίνανε μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για την ε, πιθανή μελλοντική υλοποίηση των επενδυτικών αυτών διευκολύνσεων, φαίνεται ότι ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχουν προχωρήσει πολύ περισσότερο στον τομέα των μεταφορών, ενώ από ό,τι φαίνεται υπολείπονται κάπως οι πρωτοβουλίες αυτές στον τομέα της ενέργειας ή στον τηλεπικοινωνιακό τομέα. Οι δύο τελευταίοι τομεί που ανέφερα δεν έχουν προχωρήσει τόσο πολύ όσο το μέσο των μεταφορών και αναφέρομαι πάντα στη δυνατότητα συνδυαστικών διευκολύσεων στα πλαίσια του CEF. Είναι σημαντικό λοιπόν να δοθούν τα παρέτα κίνητρα προκειμένου να προχωρήσουμε την πρωτοβουλία αυτή περισσότερο και στον τομέα τη ενέργεια και στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Πρέπει λοιπόν να επισπεύσουμε την πρωτοβουλία αυτή και για τους δύο αυτούς κλάδους, προκειμένου να καταφέρουμε να προσελκύσουμε περισσότερες ιδιωτικές επενδύσεις σε σχέδια κοινού ενδιαφέροντο στου δύο αυτού τομεί, ενέργεια και τηλεπικοινωνίε. Οι δικέ μου έχουν ως στόχο να αποσαφηνίσουν ε, καταρχά την έννοια αυτή καθεαυτήν και τι γενικότερε προθέσεις αυτής της ε, επιλογής πολιτικής και να δούμε επίση και ποιο είναι ο στόχο και ποιες οι προσδοκίε που απορρέουν από τι τροποποίησει αυτέ. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι στα πλαίσια της πρότασης για την διευκόλυνση ιδέοντα στην Ευρώπη έχουμε συντρέχους αποκλειστική αρμοδιότητα με την Επιτροπή Μεταφορών. Από κοινού δηλαδή, η δική μας Επιτροπή και η Επιτροπή Μεταφορών έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα, εν προκειμένου συντρέχους αποκλειστική αρμοδιότητα για το ζήτημα αυτό. Συνεργάστηκα λοιπόν με τον εισηγητή από την Επιτροπή Μεταφορών και ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε ένα κείμενο το οποίο θα είναι από κοινού αποδεκτό και από εμά δηλαδή και από τους συναδέλφους στην Επιτροπή Μεταφορών. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πραγματικά θέλουμε να ασκήσουμε πίεση και να επηρεάσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει το κείμενο αυτό να ετοιμαστεί το συντομότερο δυνατό, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή νομίζω ότι έχει προθεσμία μέχρι τον Μάιο ή ενδεχομένως τον Ιούνιο του 2017 για την ολοκλήρωση της πρότασης αυτής. Εν πάση περιπτώσει, στο πρώτο εξάμεινο 2017 πρέπει να ολοκληρωθεί η πρόταση. Θα ζητήσω τώρα από τους σκιώδεις συζητητές να πάρουν το λόγο, την κυρία Νούντι καταρχάς, εξ ονόματος των σοσιαλιστών. Thank you very much. Uh, ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ τον εισηγητή για την έκθεση μέχρι τώρα. Με πολλά συμφωνώ επί της ουσίας, αλλά και με τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί μέχρι τώρα. Κάνα δύο πραγματάκια θέλω να τονίσω μόνο. Το νέο προτινόμενο 274 άρθρο για το συνδυαστικό μηχανισμό. Διαφορετικά από ότι το συνδέοντας στην Ευρώπη, που είναι στο 10% του συνολικής χρηματοδότησης, το άρθρο 274 για τις τηλεπικοινωνίες δεν προτείνει ανώτατο όριο και ίσως αυτό πρέπει να το δούμε για να καταλάβουμε καλύτερα το σημείο αυτό. Δεύτερον, προφανώς πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ επιχορηγήσεων και χρηματοδοτικών μέσων και τι σημαίνουν όλα αυτά για την πορεία που θα ακολουθήσει η διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη. Προφανώς θα πρέπει να δούμε και το ποσοστό επιτυχίας των προγραμμάτων χρηματοδότησης μέχρι τώρα. Το δεύτερο σημείο που θέλω να υπογραμμίσω και το αναφέρατε και στην έκθεσή σας κι εσείς είναι το ζήτημα της απαιτούμενης διακυβέρνησης για να υπάρχει ε, απόλυτη σαφήνεια Συνδυαστικός μηχανισμός, ναι, καταλαβαίνω ε, το νόημα και το προς τα που πάει, αλλά χρειάζεται σαφής αξιολόγηση και διασφάλιση ότι τα κονδύλια χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις ε, αποφασισμένες προτεραιότητες και ότι είναι αποτελεσματικά για τις προτεραιότητες αυτές. Και αυτά τα δύο σημεία είναι πολύ σημαντικό να διασφαλιστούν. Και, όπως είπατε, και για τα σχέδια κοινού ενδιαφέροντος και ε, την παρακολούθηση της χρήσης των κονδυλίων. Αυτά είναι επίσης πολύ σημαντικά και σύμφωνο. Αυτά είναι κάποια πρώτα σχόλια και σας ευχαριστώ ξανά. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Μιλίναρ από τους φιλελευθέρους. Ευχαριστώ πρωτίστως εσάς κύριε Πρόεδρε και εισηγητά είναι καλή δουλειά. Προσβλέπω στη συνέχιση των εργασιών με τους συναδέλφους στο φάκελο αυτό. Χαιρετίζω την προσπάθεια πλούστευσης από την Κομισιόν, ε, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες Ήτρε, ε, που συνδυάζει σημαντικές αιτήσιες ε, διαδικασίες προϋπολογισμού και είναι σημαντικές οι δυνατότητες της διευκόλυνσης για την Ευρώπη και τις άλλες είναι πολύ σημαντικό και το Horizon 2020. Ο συνδυαστικός μηχανισμός είναι σημαντικό να υπάρχει, όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι. Ε, τώρα, οι γνωμοδοτικές επιτροπές, εκεί θα πρέπει να υπάρξει επικέντρωση εκεί όπου υπάρχει αρμοδιότητα. Ε, το 272-274 αντίστοιχα ε, συνέδριο στην Ευρώπη και τηλεπικοινωνίες και το 276 για το SST, για το διάστημα. Χαιρετίζω την, ε, το σχέδιο γνωμοδότησή σας και την προσπάθεια προσέλκυσης περισσότερων ιδιωτικών επενδύσεων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την πολιτική μου ομάδα. Ε, επίσης προωθείται η δυνατότητα συνδυαστικού μηχανισμού παράλληλα με μια διαδικασία διακυβέρνησης. Πιστεύω ότι οι αλλαγές που προτείνει η Κομισιόν και ο εισηγητή μας τώρα σε ό,τι αφορά τι αποκλειστικέ αρμοδιότητες της ΣΥΤΡΑ, είναι καλή λύση και όπως είπα με χαρά θα ε, συνεχίσω τη συνεργασία μου μαζί σας. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σιλικιώτης, ο επόμενο Σκιώδης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω ε, ε, Πρόεδρε και εισηγητή κύριε Πούζο για την πρόταση που έχετε καταθέσει, παρόλο που ω ομάδα, ε, ως GUNGL, έχουμε διαφορετική θέση για τους κανόνε που πρέπει να διέπουν την εφαρμογή του κανονισμού και δι για τους στόχους που πρέπει να εξυπηρετούνται. Θα έλεγα είμαστε στον αντίπαδο από ό,τι μίλησε πριν από λίγο η συνάδελφος η Μίλη Μάρα από την Άρτε. Ε, για μα, ε, βασική προτεραιότητα δεν είναι η επίτευξη τη απλούστευση όπω αναφέρεται στην έκθεση, αλλά δηλαδή η διασφάλιση τη καλύτερη αξιοποίηση των κονδυλίων του προβλησμού προς εξυπηρέτηση των αγκών και των συμφερόντων τη κοινωνία και των λαών της Ευρώπης. Επομένως, εμείς ε, δεν θα στηρίξουμε, διαφωνούμε με τη χρησιμοποίηση των διαφορών εργαλείων προτείνονται ω το προβλημό τη Ένωση να λειτουργεί ω προστασία των ιδιών των επενδυτών και να διασφαλίζει καλύτερε ηθίκε για ιδιωτικέ επενδύσει. Ιδιαίτερα όσον αφορά την πρόταση για τροπήση του κανονισμού συνδέοντα στην Ευρώπη με τη θέσπιση συνδυαστικών μηχανισμών προκειμένου να προσευχήσουν ιδιωτικέ επενδύσει, δυστυχώ το μόνο που θα επιτευχθεί, και αυτή είναι η εμπειρία που έχουμε ε, στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, είναι να αξιοποιείται ο δημόσιο πλούτο για να μειωθεί το ρίξκο για του ιδιώτε επενδυτέ. Ε, ο δικός μας ο στόχος ως GUNGL είναι να αυξηθούν τα δημόσια κονδύλια και η οικονομική στήριξη από πλευρά της Ένωσης για την άσκηση της ενεργειακής απομόνωσης, για την ανάπτυξη των απαραίτητων δημόσιων υποδομών για διασύνδεση της Ευρώπης. Αυτό έχουμε ανάγκη ε, σήμερα ε, και γι' αυτό το τοποθετούμε. Έχουμε ανάγκη δηλαδή περισσότερες δημόσιες επενδύσει, παρά ιδιωτικέ επενδύσει και προς αυτήν την κατεύθυνση θα είναι και η τροπολογίες που θα καταθήσουμε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, ε, Ευχαριστούμε πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαντάζομαι ότι ε, συμφωνεί με τα όσα είπαμε. Καταρχάς σας ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις σας συνάδελφοι. Θα απαντήσω λοιπόν εγώ τώρα γρήγορα και να κάνω και κάποιες συγκεκριμένε προτάσεις, τις οποίες μπορείτε να δείτε και στις τροπολογίες 272-274. Τώρα, διακυβέρνηση, αξιολόγηση αντικτύπου, είναι ζητήματα πολύ σημαντικά. Αν πραγματικά θέλουμε να εμβαθύνουμε και να διευρύνουμε τις δύο αυτές προτάσεις, είναι πολύ σημαντικό να προσθέσουμε κάτι σχετικό και βέβαια είμαι στη διάθεσή σας για τυχόν ε, τροπολογίες. Κυρία Μλίναρ, αναφερθήκατε στην απλούστευση. Αφού είναι πάρα πολύ σημαντικό, δεν έχουμε καταφέρει να προχωρήσουμε πάρα πολύ στο ζήτημα της απλούστευσης. Μας έχει απασχολήσει πολύ και νο... τα τελευταία 10-15 χρόνια θα έλεγα, αλλά εξακολουθεί να είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα οι προτεραιότητές μας είναι σαφείς και σε αυτές θα πρέπει να επικεντρωθούμε. Θα μπορούσε να αποτελέσει αυτό αντικείμενο συζήτηση μεταξύ της κυρίας Μλίναρ και του κυρίου Σιλικιώτη. Μια συζήτηση δηλαδή ανάμεσα στην Αγγέλικα και τον Ιωκλή. Πρέπει να καταφέρουμε να πετύχουμε την ευκταία κατάλληλη ισορροπία, γιατί χωρίς ιδιωτικές επενδύσεις δεν θα καταφέρουμε σε καμία περίπτωση να εξυπηρετήσουμε τους πολίτες μας. Θα πρέπει ακριβώς τους πολίτες αυτούς να δώσουμε τη δυνατότητα να υποφεληθούν από τις απαραίτητες ιδιωτικές επενδύσεις. Συμφωνώ λοιπόν απόλυτα μαζί σας ότι στο τέλος της όλης διαδικασίας αυτοί που θα πρέπει να αποφεληθούν είναι σίγουρα Ευρωπαίοι πολίτες, χωρίς όμως ε, ιδιωτικέ επενδύσει, αν δεν καταφέρουμε να ικανοποιήσουμε καταρχά του ιδιώτε επενδυτέ, δεν θα πετύχουμε τίποτα. Δεν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε εμεί τα πάντα από το δικό μα τον προπολογισμό, από τον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταλαβαίνετε ότι πολύ συχνά και εμείς καταβάλουμε ένα πολύ μεγάλο τίμημα από τον εθνικό και τον κοινοτικό προπολογισμό σε Ευρωπαίοι πολίτες. Είναι ζήτημα, θέλετε, αποδοτικότητα, απόδοση μάλλον των ίδιων των επενδύσεων. Και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ιδιωτικέ επενδύσει μπορεί να αποβούν ιδιαίτερα αποδοτικές. Δεν λέω ότι θα πρέπει να έχουμε κατά νου μόνο του ιδιώτε επενδυτέ και ότι αυτοί θα πρέπει να είναι το πρωταρχικό μας μέλημα. Σε καμία περίπτωση νεοκλή συμφωνώ με τι ε, παρατηρήσει σα ότι θα πρέπει να εξυπηρετήσουμε του Ευρωπαίου πολίτε. Προφανώ, συμφωνώ απόλυτα με αυτό. Απλώ λέω ότι θα πρέπει να πετύχουμε την κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα στι δύο αυτέ προσεγγίσεις. Σε κάθε περίπτωση σας ευχαριστώ πολύ για τι παρατηρήσει σα, Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσε και επικοδομητικέ. ενδεχομένω να με προκαλούν σε κάποιο βαθμό, πράγμα το οποίο μου αρέσει. Λοιπόν, να σε ενημερώσω τώρα ότι έχουμε και εδώ βέβαια προθεσμία κατάθεση τροπολογιών 9η Μαρτίου 2017. Η ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να ολοκληρώσουμε εμεί το έργο μας και να ολοκληρώσει και αυτή το έργο της μέχρι τον Ιούνιο του 2017. Επομένω δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο μπροστά μας, τέσσερις μήνες περίπου, για να ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία. Δηλαδή για να ολοκληρωθεί η πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία θα είναι έτοιμη τον, τον, τον Απρίλιο. Και στη συνέχεια βέβαια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ασχοληθεί με τα ζητήματα που άπτονται τη δική αρμοδιότητα στο πλαίσιο τη πρόταση αυτή. Α περάσουμε τώρα στο σημείο 6 τη ημερήσια διάταξη. Άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο dumping και αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρου χωρών μη μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ σημαντικό και το θέμα αυτό. Έχουμε εδώ πέρα ένα σχέδιο γνωμοδότης από τη Στάδελφο Παλώμα Λόπες Μπερμέγιο. Η ε, γνωμοδότηση αυτή απευθύνεται προς την Επιτροπή ΙΝΤΑ προκειμένου να τροποποιηθεί το σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο σχετικός κανονισμός δηλαδή, όσον αφορά τα μέτρα anti-dumping και τα μέτρα που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βέβαια ένα σχετικό ζήτημα είναι το καθεστώς οικονομίας της αγοράς, το πιθανό καθεστώς οικονομίας της αγοράς της Κίνας. Το ζήτημα αυτό μας έχει απασχολήσει πολλές φορές, έχει ανακύψει πολύ συχνά. Το 2016 η Ήτρε έχει ανταλλαγή απόψεων για το ζήτημα αυτό, παρουσία του Προέδρου Μπεντλάν και του Προέδρου της Επιτροπής Ίντα. Θυμάμαι πολύ καλά τη συζήτηση που έλαβε χώρα. Ας συνεχίσουμε λοιπόν τη συζήτηση αυτή Ας συνεχίσουμε την επεξεργασία του θέματος αυτού με την παρουσίαση που θα μας κάνει η συντάκτρια γνωμοδότησης Παλώμα Λόπεθ Μπερμέγιο, στην οποία δίνω ευθύ αμέσως το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η γνωμοδότηση της, της δικής μας Επιτροπής είναι θεμελιώδης για να καθοριστεί το μέλλον της νομοθεσίας κατά του ντάμπινγκ εντός της Ένωσης. Η αναθεώρηση αυτών των δύο κανονισμών έχει μεγάλη σημασία για το μέλλον της ευρωπαϊκής βιομηχανίας που αντιμετωπίζει ένα παγκόσμιο εμπόριο το οποίο μεταλλάσσεται πολύ γρήγορα. Για μας είναι πολύ σημαντικό πρώτα απ' όλα να μην μειώσουμε εξ αρχής τα στάνταρ προστασίας στο πλαίσιο του ΠΟΕ. Αυτό σημαίνει πρώτα απ' όλα ότι πρέπει να διατηρηθεί η δυνατότητα διάκρισης ανάμεσα στις οικονομίες αγοράς και ε, αυτό επί τη βάση των πρωτοκόλων πρόσβασης χωρών όπως η Κίνα. Επίσης σημαίνει καλύτερο καθορισμό των στρεβλώσεων τιμών που επιτρέπουν το, να ορίσουμε το dumping ως προς αυτό το σημείο. Θεωρούμε ότι η λήψη υπόψη των στρεβλώσεων όσον αφορά την φορολογία, τα χαμηλά κοινωνικά στάνταρ ή τα στάνταρ για το περιβάλλον ή το κόστος των πρώτων υλών και της ενέργειας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τη στιγμή που εξετάζεται ε, ένα πιθανό τάμπινγκ. Τέλος, θεωρούμε πως είναι σημαντικό τα συνδικάτα επίσης να μπορούν να συμμετέχουν στις έρευνες κατά του ντάμπινγκ όπου και αν αυτές γίνονται ε, με το, στο ίδιο επίπεδο με τους καταναλωτές ή τις εταιρείε, γιατί το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο στο σύνολό του είναι αυτό που θέλουμε να προστατεύσουμε με δίκαιους εμπορικούς κανόνες. Πρέπει να εγγυηθούμε τη διατήρηση του ευρωπαϊκού βιομηχανικού ιστού ως ε, ε, πυλώνα του παραγωγικού μας προτύπου, καθώς και τον κοινωνικό μας πυλώνα, τον οποίο θα πρέπει να στηρίζει το διεθνές εμπόριο και όχι να υποβαθμίζει. Γι' αυτό θα ξεκινάμε με τη βάση την πρόταση της Κομισιόν και τις ε, υποχωρήσεις που ήδη έχει κάνει το Κοινοβούλιο όσον αφορά τον εξυγχρονισμό των κανόνων αντι-dumping στην υπεράσπιση τη ευρωπαϊκή βιομηχανία. Είμαι βεβαία ότι θα έχουμε καλή συνεργασία με όλε τι πολιτικέ ομάδε ώστε να προχωρήσουμε προ αυτή την κατεύθυνση. Σα ευχαριστώ. Και εγώ σα ευχαριστώ. Συνάδελφε, και τώρα θα ακούσουμε του σκιώδεις εισηγητές μα, Ο κύριο Σαρίνη από το ΕΛΚ. Σα ευχαριστώ. Έχω την εντύπωση ότι η συγγήτρια συνέλαβε κάλλιστα το πνεύμα που εξέφρασε το Κοινοβούλιο όταν απέριψε την ευκολία με την οποία η Κομισιόν ε, θέλησε να αναγνωρίσει το καθεστώς της οικονομίας της αγοράς για την Κίνα. Εμείς είμαστε αντίθετοι για την ώρα να αναγνωρίσουμε αυτό το καθεστώς με τον τρόπο που μας προτείνεται και υπάρχει ένα πολύ λεπτό νομικό κίσης πρόβλημα γιατί στην πρόταση της Κομισιόν κατ' ουσίαν εξαφανίζεται εντό του ΠΟΕ η διάκριση ανάμεσα στις χώρες ε, που έχουν το καθεστώς και άλλες που δεν έχουν και αποφασίζει να ξεκινήσει μια πορεία σύμφωνα με την οποία εργαζόμενοι για μεμονωμένα προϊόντα μπορεί κανείς να εντοπίσει την στρέβλωση τη οποία θα πρέπει να ε, παρέμβει κανείς. Δηλαδή, ε, ε, συγκεκριμένο προϊόν, συγκεκριμένη γραμμή για το κόστος. Αυτός είναι ένας κίνδυνος τον οποίο δεν μπορούμε να διατρέξουμε και είναι ένα σφάλμα όσον αφορά την προσέγγιση στην βιομηχανική πολιτική. Υπάρχουν χώρες που ανταποκρίνονται στους κανόνες της αγοράς και άλλες που δεν ανταποκρίνονται. Και δεν μπορούμε να μετακινήσουμε ε, στις δική μας, ε, εις μας ε, το κόστος της απόδειξης. Πρέπει να ισχύει το εξής και έτσι πρέπει να παραμείνει. Μια χώρα που είναι εκτός των κανόνων της αγοράς οφείλει να αποδείξει, να φέρει το βάρος της απόδειξης ότι σέβεται τελικά τους κανόνες αγοράς. Δεν πρέπει η Κομισιόν να με λευκό επιταγή να προβαίνει ανά προϊόν σε αυτή τη διάκριση. Αυτό είναι ένα κίνδυνο στον οποίο δεν μπορεί να διατρέξει η βιομηχανία μα. Δεν είναι σαφές το νομικό πλαίσιο εντό το οποίο ορίζεται τι είναι διστρέβλωση και τι δεν είναι και δεν είναι σαφές για ποιο λόγο εμείς πρέπει να το αποδείξουμε και όχι αυτοί. Οι χώρες που πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν κάνει την κατάλληλη διαδικασία, έχουν περάσει την κατάλληλη διαδικασία για να μπορούν να θεωρηθούν οικονομίες της αγοράς. Τώρα, υπάρχει ένα τμήμα το οποίο κατά τη γνώμη μου μπορεί να μας βρει σύμφωνος και το θύμισε τώρα μόλις και η συγχύτρια. Ανάμεσα στα ένα σωρό στοιχεία που θεωρεί ότι είναι σημαντικά για να μπορούμε να εντοπίσουμε τις τριπλώσεις, μιλάει και για τη φορολογία, το θέμα της ε, ε, φορολογικής έντασης ε, σε κάποια χώρα. Γιατί είναι σωστό αυτό, γιατί σε μια χώρα όπου η φορολογία είναι πάρα πολύ χαμηλή, μπορεί όντω να συμμετέχει στη διεθνή αγορά και προβαίνει σε ένα είδο τρέβλωση. Όμω προσοχή. Προσοχή, γιατί και εμεί εδώ στην Ευρώπη, στη σήμερα ημέρα, έχουμε τέτοια κατάσταση. Έχουμε χώρε όπω η δικιά μου, όπου η φορολογική ένταση είναι τεράστια, και χώρε όπου η φορολογική ένταση είναι κοντά στο μηδέν. Είναι σωστό όμως σε ένα τέτοιο πλαίσιο μπορεί αυτό να μας οδηγήσει και να μας πούνε οι άλλοι «Μα δείτε τι κάνετε εσείς εντός της Ευρώπης, γιατί το πρόβλημα της φορολογικής εναρμόνισης δεν το έχετε λύσει ούτε εσείς στην Ευρώπη». Είναι ένα στοιχείο επί το οποίο πρέπει να δουλέψουμε, αλλά να έχουμε υπόψη μας και αυτό το στοιχείο. Ευχαριστώ και εδώ σταματώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ συνάδελφε. Βέβαια, εδώ πρέπει να δούμε και τη δική μας την εσωτερική προσέγγιση σε όλο το θέμα. Ο συνάδελφος Μαρτέν, επόμενος Κιώδης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω θα με ξεχνούσατε. Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και την Παλώμα για την πολύ καλή δουλειά που έχει κάνει και θα ήθελα να κάνω κάποιες αρχικές παρατηρήσεις. Νομίζω ότι είναι πολύ καλά το τροποποιήσαμε το χρονοδιάγραμμα, γιατί είναι πολύ σημαντικό για την Επιτροπή μας να έχει τον απαραίτητο χρόνο να ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό και να καταφέρει να καταλήξει σε μία ισχυρή τοποθέτηση για την υποστήριξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, όσον αφορά επίσης την κοινωνική, περιβαλλοντική, περιβαλλοντική, φορολογική πτυχή που θα πρέπει να είναι δίκες Νομίζω ότι θα πρέπει πραγματικά να προασπιστούμε εδώ πέρα τα συμφέροντα των 28 κρατών μελών χωρίς να δεχόμαστε τις πολιτικές που εκ των άνω θέλουν πάρα πολύ να μας επιβάλλουν. Αν λειτουργούμε με μόνο γνώμονα τις τιμές, τότε ας κλείσουμε εντελώ την Ευρώπη και ας πάμε στην Κίνα γιατί τα πάντα εκεί πέρα θα είναι εξορισμού πιο φτηνά. Ω Επιτροπή λοιπόν Βιομηχανία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και χωρί αυτή τη στιγμή να μπούμε σε μια αντιπαράθεση μεταξύ κοινοβουλευτικών επιτροπών, πράγμα το οποίο το είδαμε πριν από μερικέ εβδομάδε δυστυχώ με την Επιτροπή ΙΝΤΑ, Επιτροπή Διεθνού Εμπορίου, είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρει να ακουστεί χειρά το δικό μα το μήνυμα. Να καταφέρουμε να προασπιστούμε τη βιομηχανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχοντα μια ισότιμη και δίκαιη ένα ισότιμο και δίκαιο σύστημα ανταγωνισμού. Και αυτό ακριβώ θα ήθελα να κάνω μέσω τροπολογιών που θα υποβάλω και εγώ παράλληλα με τι τροπολογίε τη Παλώμα. Ευχαριστούμε πολύ, Πολ Ρούμπικ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Στο εμπόριο νομίζω πάντα πρέπει να προσέχουμε να υπάρχει όφελος και για τις δύο πλευρές. Απ' τη μια είναι οι καταναλωτές με που θα πρέπει να μπορούν να αγοράζουν τις ε, εισαγωγές, ε, να έχουν την απαραίτητη ε, αγοραστική δύναμη και όταν υπάρχει καλύτερη αγοραστική δύναμη μπορεί να βελτιωθούν και οι εξαγωγές και αν δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας εκεί θα μπορεί να εισπράττει περισσότερους φόρους το κράτος και πάλι θα ε, αναπτυχθεί η αγοραστική δύναμη. Είναι σημαντικό λοιπόν να ωφελήσουμε τους πολίτες μέσα από το εμπόριο. Ο προστατευτισμός ε, εδώ μόνο σε βάρος των καταναλωτών μπορεί να αποβεί. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι καλό που σκεφτόμαστε τα εμπορικά αμυντικά μέσα γιατί από τη μια πλευρά η Κομισιόν αντιμετωπίζει την Κίνα από την άλλη την Αμερική όπου ακούμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ θέλει τώρα να ε, εισαγάγει δασμούς 100% μέχρι 100% ε, δρώντας ε, στη χώρα του στα πλαίσια πολιτικής προστατευτισμού. Ε, δηλαδή θα πρέπει να πληρώνουμε 100%, θα πρέπει και οι Αμερικανοί να πληρώνουν 100% παραπάνω και επίσης θα ακριβίνουν και τα δικά τους τα προϊόντα. Θα μειωθεί λοιπόν η αγοραστική δύναμη των Αμερικανών. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να δούμε ότι την περασμένη εβδομάδα στο ε, Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου ε, κατά τα δύο τρίτητα συγκεντρώθηκαν οι υπογραφές για σωστές θελωνιακές διαδικασίες και καινούργιες ε, πρακτικές ε, η ε, απελευθέρωση θα μας δώσει και η μείωση των ρυθμίσεων θα μας ωφελήσει όλους. Η διευκόλυνση του εμπορίου, η πράξη αυτή λοιπόν που θεσπίστηκε πρέπει να εφαρμοστεί το ταχύτερο δυνατόν και στην Κίνα και τις Ηνωμένε Πολιτείες γιατί έχουμε δύο ακραίους πόλους εδώ αυτό αποτελεί μια πρόκληση για μας και για τους εργαζομένους μας και για το, το, το, τους ε, πολίτες μας. Ε, με το μέσον αυτό για το εμπόριο μπορούμε λοιπόν να αρχίσουμε μια νέα δυναμική. Ευχαριστώ. Ε, ο αντικαταστάτης κυρία Βλίναρ. Ευχαριστώ. Ελπίζω ότι οι συνάδελφοι θα κάνουν... Ελπίζω να μην μου κάνουν δύσκολες ε, ερωτήσει συνάδελφοι, γιατί θα διαβάσω τη δήλωση της κυρίας Μλίναρ. Καταρχήν ευχαριστώ τον εισηγητή, την εισηγήτρια. Ε, χαιρετίζω την πρόταση της Κομισιόν για το, νέα μεθοδολογία υπολογισμού ε, για τις εισαγωγές και τις μεθόδους ε, αντι-dumping και επιδοτήσεων κυρίως ε, με την Κίνα. Δεδομένων των σημερινών δυσκολιών, δηλαδή λήξη κάποιων διατάξεων στο πρωτόκολλο και πρόσβαση της Κίνας στον ΠΟΕ και επειδή η Κίνα ε, κάνει πολλές ε, κρατικές παρεμβάσεις ε, και στρεβλώσεις. Πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία που θα προστατεύει από τον αθέμητο ανταγωνισμό και θα σέβεται και τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του ΠΟΕ. Η αλλαγή της τωρινής μεθοδολογίας προς μια ουδέτερη προσέγγιση νομίζουμε ότι είναι σωστή πρόταση από την Κομισιόν. Δεν συμφωνεί με τη θέση της εισηγήτριας να υπάρξει αναφορά σε καθεστώς ε, οικονομίας αγοράς ή όχι για τα μέλη του ΠΟΕ είναι σημαντικό για την προστα... πρέπει να προστατεύσουμε τη βιομηχανία αλλά χωρίς προστατευτισμό. Την πρόταση θα πρέπει να τη δούμε στο ευρύτερο πλαίσιο του στόχου να ενισχύσουμε ε, ένα σύστημα εμπορίου που θα στηρίζεται σε κανόνες. Τέλος, υπάρχουν και ορισμένα ανοιχτά ερωτήματα που πρέπει να δούμε, που αφορούν ιδιαίτερα το ρόλο της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και την ενδεχόμενη αντιστροφή του βάρους των αποδείξεων και την συνέπεια των εκθέσεων αναχώρα που θα ε, ε, καταρτίζει η Κομισιόν. Θα πρέπει να ε, τα δούμε όλα αυτά στα πλαίσια μιας συνεργασίας στην οποία προσβλέπω με τους αγαπητούς συναδέλφους. Ευχαριστώ πολύ. Ο συνάδελφος Χόφερ για τους Πρασίνους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαιρετίζουμε την πρόταση της Κομισιόν θεωρούμε ότι πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση. Όμως ακόμα υπολείπεται σε σχέση με τα κριτήρια που είχε θέσει το Κοινοβούλιο. Συμφωνώ με τους συναδέλφους που είπαν, όπως και ο συνάδελφος Φέντερ πριν από λίγο, που αντικατέστησε την συνάδελφό του, Συμφωνώ με εκείνους που λένε ότι έχουμε ε, ένα διπλό σετ κριτηρίων να εφαρμόσουμε. Η λύση που θα βρούμε θα πρέπει να είναι συμβατή με τον ΠΟΕ, αλλά πρέπει επίσης να μας επιτρέπει να ε, ε, εφαρμόζουμε συστήματα άμυνα στο εμπόριο. Αλλιώς ο αθε... μπορεί να αντιμετωπίσουμε ε, προβλήματα λόγω αθέμη ανταγωνισμού. Δεν πιστεύω ότι σε αυτό το πλαίσιο χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε ρητά τον όρο καθεστώς οικονομίας αγοράς ή όχι. Νομίζω ότι καλό θα ήταν να αποφύγουμε αυτούς τους όρους. Όμως δεν μπορούμε να ξαναγυρίσουμε στον συνήθι τρόπο εφαρμογής της ε, μεθοδολογίας, της στάνταρ μεθοδολογίας. Πρέπει να βρούμε μια ειδική μεθοδολογία που θα μας επιτρέπει αποτελεσματική άμυνα απέναντι στον αθέμητο ανταγωνισμό. Η μετατόπιση του βάρους των αποδείξεων στην ευρωπαϊκή πλευρά είναι πιο αδύναμη από αυτή που θα ήθελα εγώ. Δεν βλέπω λόγο γιατί να μην κάνουμε και εμείς το ίδιο όπως οι Αμερικανοί που επέμειναν το βάρος των αποδείξεων να βρίσκεται στο άλλο μέρος. Αν όμως η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη δεν τολμούν να σηκώσουν το ειδικό τους βάρος υπέρ μιας τέτοιας επιλογής, τότε τουλάχιστον η διάταξη που θα θέσουν επιτάπητος θα πρέπει να γίνει πιο στιβαρή. Η γλώσσα που επιλέγουμε τώρα δεν, ε, δεν διασφαλίζει ότι η έκθεση θα ισχύει παντού, όποτε θα χρειάζεται. Αν η Κομισιόν δεν ε, παρουσιάσει ένα σύστημα αναφοράς και εκθέσεων. Δεν έχουμε βάση να αποδείξουμε ότι οι πρακτικές που χρησιμοποιεί η άλλη πλευρά είναι αθέμητες και ότι υπάρχει dumping. Πρέπει να το επεξεργαστούμε καλύτερα αυτό. Δεύτερο πρόβλημα που βλέπω. Σύμφωνα με το Κινέζικο Πρωτόκολλο Προσχώρησης, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και αμυντικά μέσα κατά των επιδοτήσεων και αυτά δεν προσδιορίζονται, ε, δεν περιορίζονται χρονικά, δεν λήγουν. Η Κομισιόν δεν το λαμβάνει υπόψη της αυτό. Ακόμα φαίνεται να υπαναχωρεί σε σχέση με την υφιστάμενη νομική βάση για την ε, χρησιμοποίηση τέτοιων μέσων στο μέλλον. Αυτό δεν είναι καλό, είναι υπερβολικά αμυντικό και πρέπει να το βελτιώσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Μπορέλη, εξ ονόματος της CFDD. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι οικονομικές επιπτώσεις και βιομηχανικές επιπτώσεις της νομοθετικής αυτής πρότασης είναι γνωστές σε όλους. Εμείς βλέπουμε ότι υπάρχει ένας κίνδυνος για πάρα πολλούς βιομηχανικούς τομείς στην Ευρώπη με επιζήμιες συνέπειες από κοινωνικής πλευράς και όσον αφορά την ευρωπαϊκή τεχνογνωσία. Έχουμε από την άλλη την τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπου, λέμε ότι, όπου λέει ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε πάρα πολύ γρήγορα και ενδεχομένως βέβαια να βρεθούμε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση στα πλαίσια του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίας. Γι' αυτό μας λέει, ότι η Ευρωπαϊκή, μας λέει Επιτροπή ότι θα πρέπει να καταλήξουμε σε έναν ουδέτερο κανονισμό που να μας επιτρέψει να περαμηθούμε της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περίπτωση διαφορών. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο ορισμό όσον αφορά το ζήτημα της τρέβλωσης αν πούμε τώρα όμως στην ουσία της γνωμοδότησης της δική μας Επιτροπής, καταρχάς να ευχαριστήσω την ε, εισηγήτρια, η οποία προσπάθησε να εξορροπήσει κάπως την πρότασή μας και κάνει μια διάκριση ανάμεσα σε καθεστώς ή μη οικονομίας της αγοράς. Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό σε σχέση με τους εμπορικούς μας εταίρους και με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Ένας από τους παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν στρέβλωση ακόμα και στον τομέα της ενέργειας είναι ότι δεν έχουμε συγκεκριμένες συνθήκες και προϋποθέσεις όσον αφορά το περιβάλλον, την κοινωνία, τη φορολογία. Ξέρετε ότι υπάρχουν κάποιες χώρες οι οποίες κινδυνεύουν περισσότερο. Είναι σημαντικό επίσης να λάβουμε υπόψη μας τη συμβολή όλων των διαφορεμένων μερών. Θεωρώ ότι θα πρέπει να ενισχυθούν οι αρχικές αυτές προτάσεις της συγγήτριας θα πρέπει να αναφερθούμε πιο συγκεκριμένα στις στρεβλώσεις. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να, γίν να ακολουθήσουμε αυτή την ξεκάθαρη διαφορά, διαφοροποίηση που υπάρχει ανάμεσα στο καθεστώς σημεί της οικονομίας της αγοράς, στο, στον κανονισμο αντιντάμπινγκ anti-dumping αυτή τη στιγμή, αλλά και στην προσχώρηση, στο πρωτόκολλο προσχώρησης, δεν γίνεται αυτή η σημαντική διάκριση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν στα πλαίσια της αγοράς να χρησιμοποιούνται τα πέντε αυτά κριτήρια. Κατά αυτόν τον τρόπο το βάρος της απόδειξης θα βαρύνει τελικά αυτόν ο οποίος ε, τηρεί ή δεν τηρεί τα πέντε αυτά κριτήρια για συμμετοχή στην οικονομία της αγοράς. Πραγματικά αυτή τη στιγμή θέλουμε να ε, εισάγουμε την έννοια αυτή της στρέβλωσης όπως παρουσιάζεται στην πρόταση κανονισμού, η οποία έννοια παραμένει πάρα πολύ ασαφή αυτή τη στιγμή. Και τι θα κάνουμε απέναντι στην Κίνα, για παράδειγμα. Καταλαβαίνετε ότι για τι ευρωπαϊκέ βιομηχανίε θα ήταν αδύνατο να εφαρμόσουμε την έννοια αυτή και τα κριτήρια τα οποία περιλαμβάνονται. Και επίση τι θα κάνουμε αυτή τη στιγμή με του διεθνεί εταίρους μα, αλλά και του ίδιου του εργαζόμενου στην Ευρωπαϊκή Ένωση που περιμένουν μια στιβαρή τοποθέτηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να προασπίσουμε την απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Βιομηχανία αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να είναι η προτεραιότητά μας και όχι να υιοθετήσουμε τελικά θέσεις οι οποίες θα είναι πάρα πολύ ασαφείς από νομικής πλευράς. Πραγματικά δεν γνωρίζουμε αν εφαρμοστεί η πρόταση αυτή ποια θα είναι η έκβαση για την Ευρωπαϊκή Ένωση αν εμπλακεί σε νομικές δικαστικές διαφορές με άλλες χώρες όπως για παράδειγμα με την Κίνα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Πασίωρ από το Άρνης και ο δισηγητής για αυτή την ομάδα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη που ζητώ τόσο απότομα τον λόγο. Είχα χάσει το τρένο μου, χρειάστηκε να κάνουμε παράκαμψη για να φτάσω εδώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε το λόγο. Να ευχαριστήσω την συντάκτρια γνωμοδότησης από την ΚΟΕ Χαίρομαι πάρα πολύ που αναγνωρίζει ότι το τομέα ενέργεια είναι πάρα πολύ σημαντικό για το διεθνέ εμπόριο και ιδίω μετέρου εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Ω Ευρωβουλευτή όμω που προέρχεται από το Yorkshire, μια περιοχή τη Μεγάλη Βρετανία που πραγματικά έχει πληγεί από την κρίση στη Χαλιβουργία, γνωρίζω πραγματικά ότι μπορεί να προκληθούν πάρα πολλά προβλήματα στο βιομηχανικό τομέα. Προκειμένου λοιπόν να καταφέρω να συμβάλλω σε μια πλήρη και ευρία γνωμοδότηση για ένα ζήτημα το οποίο είναι τόσο πολιτικό όσο και τεχνικό, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε όλοι να κατανοήσουμε καλύτερα κάποια επιμέρου ζητήματα. Θα μπορούσαμε για παράδειγμα να δούμε πώς έχουν τα πράγματα και συζητήσεις αυτή τη στιγμή όσον αφορά την ε, στάση της ε, Κίνας απέναντι στους κανόνες anti-dumping σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε επίπεδο παγκόσμιου οργανισμού εμπορίου. Μολονότι θεωρούμε ότι θα πρέπει να εξυγχρονιστούν τα εμπορικά αμυντικά μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να διασφαλίσουμε παράλληλα ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τον υπολογισμό των περιθωρίων anti-dumping θα προωθήσουν την ελεύθερη αγορά και θα τηρήσουν τις προϋποθέσεις ελεύθερης αγοράς και θα πρέπει αυτό να ληφθεί υπόψη σε σχέση με την στάση που θα κρατήσουμε απέναντι στην Κίνα. Οι αθέμητες εμπορικές πρακτικές όπως το dumping που αποτελούν πολλές φορές αποτέλεσμα της παρέμβασης των κρατών μελών στη ελεύθερη αγορά είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αποτραπεί. Θα πρέπει σε όλα τα επίπεδα, σε όλη την ε, αλυσίδα εφοδιασμού, να μην έχουμε μια παρεμβατική στάση των κρατών μελών, όπου θα πρέπει και αυτά να τηρούν τους κανόνες ελεύθερης αγοράς. Επομένως, αντιτιθήμεθα σε οτιδήποτε υπερβαίνει τη δημιουργία ενός ισότιμου, ισότιμου πεδίου ανταγωνισμού και κάτι το οποίο θα ε, συνέβαλε τελικά στο να δημιουργηθούν κάποιοι προστατευόμενοι εμπορικοί τομείς στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόεδρος. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος άλλος το λόγο, αγαπητοί συνάδελφοι. Δεν νομίζω. Ο κύριος Μιούλερ από την Γενική Διεύθυνση Εμπορίου προσωπώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Thank you. Thank you, Mr. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και το συγγνώμη που έφτασα λίγο καθυστερημένα. και έτσι έπεσα στη μέση της συζήτησης. Η Κομισιόν θα ήθελα να ευχαριστήσει την εισηγήτρια για την έκθεση που έκανε ε, και για την ε, καλή της ε, εξαιρετική της εργασία. Η Κομισιόν θα ήθελε να τονίσει ότι τρία από τα τέσσερα στοιχεία της πρότασης καταρχάς ήδη καλύπτονται από την πρόταση της Κομισιόν και ήδη έχουμε μιλήσει για αυτές τις ιδέες. Το πρώτο σημείο το οποίο τόνισε η συγγήτρια είναι ο ορισμός της σημαντικής στρέφλωσης, ότι δηλαδή αυτή θα πρέπει να καλύπτει και τη φορολογία, το κόστος στο περιβάλλον και το κοινωνικό κόστος. Το τρίτο αφορά τους εργαζόμενους και την εκπροσώπηση των συνδικάτων και το τελευταίο αφορά την αντιμετώπιση χωρών ε, χωρίς οικονομία της αγοράς όπως το, η Κίνα και το ε, Βιετνάμ. Όσον αφορά την ενέργεια, το κόστος της ενέργειας και το τι σημαίνει αυτό, η Κομισιόν τονίζει ότι η ενέργεια είναι σημαντικό στο ε, συνιστός της παραγωγής και άρα αυτόματα αναλύεται στον καθορισμό της τρέβλωσης. εργασιακά, περιβάλλον, φορολογία επίσης εξετάζονται διότι το εργατικό κόστος καλύπτεται, είναι σημαντικό κόστος παραγωγής. Ε, το θέμα της φορολογίας καλύπτεται εάν είναι κάποιο μέτρο που δημιουργεί και προκαλεί στρέβλωση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η φόρη εξαγωγών, που είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα στρέβλωσης και καλύπτεται. Τώρα, το θέμα περιβαλλοντικών προτύπων είναι πιο ευαίσθητο, γιατί δεν υπάρχει συμφωνημένο κατάλογος σε εθνικό επίπεδο που θα αναφερόταν σε αυτά τα πρότυπα. Εκεί δεν υπάρχει συμφωνημένο κατάλογος. Η Κομισιόν θέλει να τονίσει επίση ότι στη μεθοδολογία του ντάμπινγκ, όπως έχει σήμερα, ε, υπάρχουν ε, τα εργατικά και περιβαλλοντικά κόστη ε, και το περιθώριο βλάβης. Και αυτό το έχει υπολογίσει η Κομισιόν. Δηλαδή το κόστος παραγωγής ευρωπαϊκής βιομηχανίας που περιλαμβάνει και τα κόστη για την ευρωπαϊκή βιομηχανία όταν εφαρμόζει τα πρότυπα για το τομέα της εργασίας και το περιβάλλον. Τώρα, τρίτο σημείο της εισηγήτριας, τα συμφέροντα των εργαζομένων ε, τα συνδικάτα και οι έρευνες για την ε, εμπορική άμυνα. Ε, τα θέματα αυτά για τα συνδικαλιστικά δεν καλύπτονται από την πρόταση. Ε, το, το, και, συγγνώμη, όχι το, ε, η, δοκιμασία, η δοκιμή για τα συμφέροντα της Ένωσης. Αυτό είναι κομμάτι του παράλληλου εγχειρήματο εξυγχρονισμού. Ε, αυτό το θέμα δηλαδή καλύπτεται εκεί. Και ε, υπάρχουν θα, τώρα, θα αρχίσουν σύντομα, τέλος Μαρτίου, τριμερείς διάλογοι για αυτό το θέμα. Ας δούμε τώρα το τελευταίο, αλλά πολύ σημαντικό θέμα. Δηλαδή η αντιμετώπιση των μελών του ΠΟΕ που δεν είναι χώρες οικονομίας της αγοράς. Για την Κομισιόν, αυτό είναι το προβληματικό κομμάτι της πρότασης που αναφέρεται στον, στο άρθρο 27 του βασικού κανονισμού. Η Κομισιόν πιστεύει ότι δεν είναι καλή ιδέα να ακολουθήσουμε την πρόταση εκεί. Ουσιαστικά η πρόταση σημαίνει ότι δεν πρέπει να αλλάξουμε τίποτα ε, για τις χώρες που δεν είναι οικονομίες της αγοράς και είναι στον ΠΟΕ. Ο λόγος της πρότασης αυτής από την Κομισιόν είναι να έχουμε ένα μέσο ουδέτερο σε σχέση με τις χώρες και να μην γίνεται διαφοροποίηση μεταξύ ε, χωρών του ΠΟΕ που έχουν οικονομία της αγοράς και τις άλλες. Η Κομισιόν πιστεύει ότι η νομική διάκριση για τα μέλη του ΠΟΕ δεν ε, αντιμετωπίζει αποτελεσματικά το θέμα των στρεβλώσεων που βρίσκονται στη ρίζα του αθέμητου, του, εμπορίου. Ε, επίσης, ε, η Κομισιόν προσθέτει ότι η πρόταση ξεκαθαρίζει ότι δεν χορηγεί σε καμία χώρα καθεστώς οικονομία τη Ε, Σε σχέση με αυτό το τελευταίο, τις αλλαγές στο άρθρο 27, αυτό δεν πρέπει να ε, μας κάνει να ξεχάσουμε το καλό έργο ε, που έχει επιτελεστεί στα πλαίσια της έκθεσης αυτής. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, η συγγήτρια, η κυρία Λόπες Μπερμέχο. Do you want to add Έχετε κάτι. Κάτι. Α, ο κύριος Μαρτέν θέλει κάτι να προσθέσει πριν να ε, κλείσει η συγγήτρια. Ναι. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, λυπούμε που παίρνω το λόγο πριν από την κυρία Βερμέχο Λόπες, αλλά απλά επειδή δεν θέλω να γίνει τώρα η συζήτηση, δεν είναι η κατάλληλη στιγμή σας είπα θα υποβάλω κάποιες τροπολογίες, αλλά αντίθετα θα ήθελα να αντιδράσω σε κάτι που υπόθηκε και να πω ότι είναι αντίθετο αυτό που είπε, ότι δεν υπάρχει λέει διεθνές ε, έγγραφο που να επιτρέπει την ανιχνευσιμότητα για τα περιβαλλοντικά ζητήματα, όμως για το διοξείδιο του άνθρακα, ας πούμε για το διοξείδιο του άνθρακα και επιτρέψατε μου να σας πω ότι σε όλες τις επιχειρήσεις του κόσμου είτε είναι στην, αγορά, στην οικονομία της αγοράς είτε όχι, απαιτείται από τον, από τον πελάτη. Υπάρχει τεχνικό, ε, τεχ, τεχνικό όπου υπάρχουν όλα τα στοιχεία. Πώς φτιάχτηκε, από ποιον, ποιος πώς, ε, ποια ενέργεια, πόση ενέργεια καταναλώθηκε, αν υπήρξε κάποιο... Ε, περιστατικό στη διαδικασία παραγωγής και λέει ας πούμε φτάνει να γράψει κανείς χρησιμοποιήθηκε τόσο διοξίδιο του άνθρακα για να, για την παραγωγή του τάδε προϊόντος. Υπάρχει ήδη διεθνή ε, τεχνική λοιπόν, αλλά πρέπει να υπάρχει και η πολιτική βούληση ώστε να αναγράφεται αυτό στο τεχνικό δελτίο κάθε προϊόντος. Ευχαριστώ. Η συγχύτρια. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συζήτηση αυτή. Είναι προφανές ότι όλοι θέλουμε να προχωρήσουμε σε καλύτερη ε, ε, εφαρμογή των γενικών κανόνων του ΠΟΕ ε, και όσον αφορά την τήρηση των δεσμεύσεων που έχουμε αναλάβει στο παρελθόν. Ε, και επίσης θέλουμε εμπορικούς κανόνες που να επιτρέπουν την άνθηση των, ε, των επιχειρήσεών μας και θα ενισχύουν την οικονομία μας. Αυτό το νόημα έχει η πρότασή μας και αυτό, μέσα σε αυτό το πνεύμα την υλοποιήσαμε και δεν θέλουμε να κάνουμε καμιά επιλογή όχι θέλουμε να έχουμε περισσότερες επιλογές για τη βιομηχανία μας και όχι λιγότερες όσον αφορά το κριτήριο της, ε, της ε, οικονομίας της αγοράς. Θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Ε, θα δούμε τα υπόλοιπα θέματα και δεν αμφιβάλλω ότι η συζήτηση για τις τροπολογίες θα μας δώσει και την ευκαιρία την καρποφόρα ώστε να συνεχίσουμε την πρόοδο και να φτάσουμε σε μια συμφωνία στο θέμα αυτό και σας ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ και εγώ πολύ. Προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών η 15η Μαρτίου 2017. Μία το απόγευμα. Μία το μεσημέρι. Δηλαδή μια ώρα περισσότερο από ό,τι ήθιστε. Συνήθως είναι 12 το μεσημέρι. Έχουμε πολύ χρόνο. Να θυμίσω 9 το πρωί έχουμε συντονιστές και όλοι μαζί ξανά συνεδριάζουμε στις 10. Το απόγευμα όμως είναι πολύ σημαντικό να θυμίσουμε ότι αύριο ξεκινάμε 4 ε, παρατέταρτο και σε άλλη αίθουσα. 5 Β01 είναι στο ίδιο κτίριο στον 5ο όροφο. 5Β01 αύριο στι 9 ε, συντονιστέ συντονιστές στις 10 ψηφοφορίε. Ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε αύριο. That's